Chers collègues, bonjour. Je vous propose de, de commencer. Πάμε, ξεκινάμε. Κατανοώ βέβαια όλους αυτούς που έχουν να αντιμετωπίσουν το σημείο 22 ότι μπορεί να μείνει ακόμα παρόντες μαζί μας. Έχουμε όμως την συγγήτρια την κυρία Αρκίν και ορισμένους σκιώδης. Προτείνω λοιπόν να επανέλθουμε στις εργασίες μας. Στο σημείο 22 δίνω το λόγο στην κυρία Χάρκιν σε σχέση με την έκθεση πρωτοβουλίας της «Αναγνώριση και αξιοποίηση των εθελοντικών ενεργειών διαμεθοριακού χαρακτήρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ψέματα δεν είναι έκθεση πρωτοβουλίας, αλλά γνωμοδότηση για την Επιτροπή Πολιτισμού. Και σήμερα εξετάζουμε αυτό το σχέδιο Έχετε το λόγο κύριε Χαρκίν. Είναι... Μετά την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινηθήκαμε που προωθεί ε, τις δραστηριότητες αυτές τις συνοριακές και ακολουθεί και το έτος εθελοντισμού το 2011. Ένα από τα πρώτα που αναφέρω και που αναφέρεται και σε αυτούς περί θελοντισμού είναι ότι ο θελοντισμός δεν θα πρέπει να ε, υποκαθιστά την ε, αμοιβόμενη εργασία διότι πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Κυρίως όταν περικόπτονται υπηρεσίε και η διαχωριστική γραμμή είναι λεπτή και δύσκολο να καθοριστεί καμιά φορά μεταξύ των δύο. Ε, είναι σημαντικό να αναφέρεται στην αρχή αυτό το πράγμα, το ξεκαθαρίζουμε. Στο 4, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 να αναπτύξει υποστηρίξει πρωτοβουλίε, ούτω ώστε να συμβάλλει ο θελοντισμό σε ευφυή, βιώσιμη και ενταξιακή ανάπτυξη. Ε, όσον αφορά την ευφυή ανάπτυξη τώρα, θα πρέπει να υπογραμμίζουμε διάφορα προγράμματα όπως η νεολαία κινήση, όπου αναγνωρίζεται η ανεπίσημη ε, μάθηση και βελτιώνεται έτσι η απασχολησιμότητα στον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πολλοί εθελοντές συμμετέχουν σε προγράμματα για την καταπολέμηση αλλαγής του κλίματος και άλλα. Και ενταξιακή ανάπτυξη, ο εθελοντισμός προωθεί ε, την ένταξη για να βελτιώνονται ευκαιρίες που δίνονται. Όσον αφορά το διαβατήριο το ευρωπαϊκό για τις δεξιότητες, έχουμε το Europass τώρα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τη ΣΕΝΤΕΦΟΠ θέλουν να ετοιμάσουν νέο έγγραφο. Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων που και αυτό θα καταγράφει την ανεπίσημη εκμάθηση. Ε, κάτι που δεν πιστοποιείται κατά διάρκεια εθελοντικών εργασιών. Σημείο 6. Ζητώ επαρκή χρηματοδότηση. Εκεί αναφέρομαι στο πρόγραμμα GrantFig που υποστηρίζει ηλικιωμένους ε, εθελοντές. και αναφέρεται ότι υπάρχει κίνδυνος περικοπής αυτού του προγράμματος. Στο σημείο 7 για τις συνοριακές εργασίες υπάρχουν κάποιες ερωτήσει από τους συναδέλφους. Το είδα σε κάνα δύο έγγραφα αυτό. Εάν οι εθελοντές θέλουν να πρέπει να περάσουν τα σύνορα, καμιά φορά είναι πιο εύκολο αυτό να γίνεται προ γειτονική χώρα. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν ε, ομοιότητες στη γλώσσα, στον πολιτισμό και το κόστος δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι ένα πρώτο βήμα. Μερικοί πάνε από τη Ρώμη στο Όσλο για εθελοντικέ εργασίε. Οι πιο ηλικιωμένοι συνήθω απλώ θέλουν να περάσουν τα σύνορα και να πάνε σε μια γειτονική χώρα. για να ενθαρρύνουμε διασυνοριακό εθελοντισμό, ίσω θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με μικρά βήματα. Τώρα, όσον αφορά κάποια έγγραφα που εξέτασα, είδα ότι υπάρχουν διάφοροι φραγμοί και όρια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν θέλουν να κινηθούν στα πίστα εθελοντισμού και να πάνε σε άλλες χώρες. Όταν διαμένουν σε μια χώρα και θα ταξιδέψουν να πάνε σε μια άλλη. Ε, πρέπει να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, τα εμπόδια, ούτω ώστε να μην υπάρχουν φραγμοί όσον αφορά τον ε, εθελοντισμό. 9. Το έχω αναφέρει ξανά να χρησιμοποιώ ε, η χρήση του χρόνου εθελοντισμού για χρηματοδότηση διάφορων ε, ευρωπαϊκών ε, προγραμμάτων. Είναι ένα κίνητρο για να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα οι εθελοντές. Στο σημείο 10 ζητώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θαρρύνει τα κράτη-μέλη να θετήσουν το εγχειρίδιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για τον εθελοντισμό. Πολλά κράτη-μέλη έχουν εγκρίνει αυτό το εγχειρίδιο και άλλα είναι καθοδόν. Αν ίσχυε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, θα είχαμε συγκρίσιμα στοιχεία, αξιόπιστα, τα οποία τα χρειαζόμαστε για τις πολιτικές που διαμορφώνουμε. Αυτά, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξέρω τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι και αν τυχόν έχουν άλλες ιδέες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Αντικαθιστώ την κυρία Μπερές για λίγο. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Η κυρία Ράπτη τώρα και ο κύριος Έλμερ Κυρία Ράπτη τώρα. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την ανάληψη των καθηκόντων σας και τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Ε, να ευχαριστήσω την κυρία Χάρκινγκ για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η εμπειρία της είναι πάντα πολύτιμη και αποτυπώνεται πάντα στις εισηγήσει της, είτε για εκθέσεις είτε για γνωμοδοτήσεις. Ε, δύο σημεία ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω. Ε, αφορούν το σημείο 2 και το σημείο 3. Στο σημείο 3 διαβάζω ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, ενώ παράλληλα συντείνει στην επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Ε, θα ήθελα ίσως να σκεφτούμε το γεγονός ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει, το λέω περιφραστικά, το λέω με πολλά λόγια, μπορούμε να δούμε πώς ε, μπορούμε να το εντάξουμε, αν η κυρία Χάρκιν συμφωνεί, μέσα στη γνωμοδότηση, ο εθελοντισμός συμβάλλει και στο να αισθάνονται οι άνθρωποι χρήσιμοι. Και μιλάω κυρίως για ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν πάρει σύνταξη, αλλά μπορούν να είναι ενεργοί, μπορούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, είτε για ανθρώπους οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν να μπουν μέσα στην αγορά εργασίας, αλλά έχουν γνώσεις και προσόντα που μπορούν να είναι χρήσιμα στον εθελοντισμό. Και το σημείο 3 στο οποίο αναφέρεται ότι ο εθελοντισμός δεν πρέπει να υποκαθιστά την αμοιβόμενη εργασία. Εγώ θα πρότεινα ότι ο εθελοντισμός παράλληλα δεν θα πρέπει να υποκαθιστά και το κοινωνικό κράτος στις υποχρεώσεις του. Αυτά είναι τα δύο σημεία που έχω στο μυαλό μου και που είμαι ε, ανοιχτή βεβαίως ε, εάν και η κυρία Χάρκινγκ νομίζει ότι αξίζουν τον κόπο να μπουν στη γνωμοδότηση ενδεχομένως και να συνυπογράψουμε ε, κάποιες τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, καλή δουλειά κυρία Χάρκινγκ και στη συνέχεια. Εντάξει, Ευχαριστώ. Ακούω την συζήτηση αυτή και πρέπει να σας πω ότι φτάνει στα όρια του σουρεαλισμού. Τι να σκεφτώ τον Έρωνα που έπαιζε βιολίδι ενώ και εγώ ήταν η Ρώμη, τη δεξίωση στον Τιτανικό όταν βυθιζόταν το πλοίο, τι να σας πω. Είναι εδώ μια υπαρξιακή κρίση φαίνεται στην Ευρωζώνη και την Ένωση. Και εμείς μιλάμε για διαμεθοριακό εθελοντισμό. Τέσσερα εκατομμύρια εκλογής μου στην ε, Βρετανία. Κανείς δεν μου είπε θέλω εθελοντισμό αλλά σε άλλη χώρα. Υπάρχει η ζήτηση για αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε γι' αυτό. Γνωρίζω ότι υπάρχουν εθελοντές για να πάνε να κάνουν κάτι σε χώρες του τρίτου κόσμου για να οικοδομηθεί ένα σχολείο ή μια κλινική στην Αφρική. Ακούσαμε ότι κάποιος ζήτησε λέει να πάει εθελοντής από την Ιταλία στο Όσλο. Μα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ποιο Ιταλό ζητάει να πάει στο Όσλο. Οι εθελοντές ζητούν συνήθως να βοηθήσουν την κοινότητά του την τοπική. Και αν θέλετε πέστε με απλοϊκό, αλλά εγώ νόμιζα ότι ο εθελοντισμός ήταν εθελοντικός. Τώρα βλέπουμε ότι δημιουργείται ολόκληρη πολύπλοκη γραφειοκρατική ευρωπαϊκή δομή για να διευθετήσει τα του εθελοντισμού. Αυτά μου φαίνονται πολύ περίεργα και πάλι εξ ονόματος των τεσσάρων εκατομμυρίων εκλογέων μου αναρωτιέμαι αυτά που ακούμε έχουν καμία επίπτωση στη ζωή του κόσμου που εκπροσωπούμε. Ακούσαμε για το πρόγραμμα Youth on the Move. Εγώ δεν άκουσα κανέναν στην περιφέρειά μου που να το έχει καν ακούσει. Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων. Ποιος έχει ακούσει ποτέ τίποτα γι' αυτό. Μήπως υπάρχει μόνο εδώ μέσα για να αυτοικανοποιούμαστε. Και άλλο παράδειγμα που το είπαμε χθες. Το ευρωπαϊκό λέει έτος ενεργούς γυράνσεως. Τι θα πει αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι 60 χρονών και ίσως είμαι υπόδειγμα ενεργούς γυράνσεως, αλλά δεν ξέρω κανέναν από, τους 4, από τα 4 αυτά εκατομμύρια που να έχει βοηθηθεί από καμία πτυχή αυτού του προγράμματος ανεργούς γυράνσεως. Εγώ είμαι εδώ 12,5 χρόνια και έχω την εντύπωση ότι δημιουργούμε θέσεις εργασίας για τους εαυτούς μας και μιλάμε μεταξύ μας για πράγματα που δεν έχουν απολύτως καμία σημασία έξω από αυτούς τους τέσσερις τείχους. Ευχαριστούμε κύριε Έλμερ. Ορισμένοι συνάδελφοι θα απαντήσουν φαντάζομαι στα ερωτήματα που θέσατε. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε όμως και ψηφοφορίες. Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους να βιαστούν. Μιλήσατε αρκετά προκλητικά, θα μιλήσουν και οι άλλοι λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό που άκουσα ε, δείχνουν διαφορές μεταξύ περιφερειών. Κάποια από αυτά που υπόθηκαν ισχύουν. Ξέρω και άλλα όχι. Ήρθαν κάποιοι από Γερμανία για να πάνε στο Ανατολικό Λονδίνο για εθελοντικές εργασίες. Ενδιαφέρονται ο κόσμος για διασυνοριακό εθελοντισμό. Ίσως όχι σε μαζική κλίμακα, αλλά ενδιαφέρονται. Και κάποια από τα θέματα που αναφέρονται, όπως σημείο 8 για την ασφάλεια δικαίου, είναι αρκετά σημαντικά στο πλαίσιο αυτό. Πώς εφαρμόζονται η κοινωνική ασφάλιση, η ασφάλιση κλπ και πώς επηρεάζονται. Και αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που θίγονται. Δύο-τρία σημεία θα ήθελα να προσθεθούν. Είναι έξοχη η γνωμοδότηση. Καλύπτει τα βασικά σημεία. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα απ' όλα το θέμα για την υποστήριξη των εργοδοτών για τους εθελοντές είναι μεγάλο θέμα σε αρκετά κράτη-μέλη και αφορά και την εταιρική ευθύνη, κοινωνική ευθύνη των εταιριών. Και ίσως κάτι θα έπρεπε να πούμε πάνω σε αυτό και θα ήθελα να υποβάλω σχετική σύντομη τροπολογία. Και πώς ενθαρρύνουμε ποικιλομορφία όσον αφορά τον θελοντισμό. Αναφέρθηκε κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο που καλύπτει συγκεκριμένο τομέα, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. αυτές τις μικρές, τις δύο μικρές προστίκες θα ήθελα να κάνω σε μια γνωμοδότηση την οποία θεωρώ έξοχη. Ευχαριστώ Τζιν. Τόμας Μαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητή μου, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω σε αυτή την επίσημη θέση. Ευχαριστώ πολύ τη Μαριάν. Η Μαριάν ήταν δασκάλα Άρα μπορεί να τα λέει καθαρά τα πράγματα με εκπαιδευτικό τρόπο και μας έχει δώσει πολλές εκθέσεις τέτοιου είδους. Τώρα να απευθυνθώ προς τον Ρότζερ Χέλμερ. Ρότζερ, χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να είναι θελοντές, που σκέφτονται τι μπορούν να κάνουν για τη χώρα, τι μπορούν να κάνουν για την κοινωνία, τι μπορούν να κάνουν παραπάνω χωρίς να ζητούν χρήματα γι' αυτό. Είναι άνθρωποι που λένε θέλω να κάνω κάποια συνεισφορά. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο να το έχουμε αυτό στην ε, κοινωνία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ε, συμμετέχουν στον εθελοντισμό και στο έτος εθελοντισμού και πρέπει να ανοίξουμε τις δυνατότητες που θα έχουν. Δεύτερον, η ενεργός γύρανση το 2010 συνέταξα μια έκθεση αυτή την Επιτροπή όσον αφορά την δικαιοσύνη ε, μεταξύ γενεών. Και είχα ρωτήσει τότε, είχα ζητήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει αυτό το έτος για ενεργό γύρανση και το έχουμε τώρα. Και θα γίνουν διάφορα πράγματα το 2012. Τι σημαίνει. Κάποιος σαν τον Έλμαρ που είναι πάντα δραστήριος και προκλητικός δεν είναι ηλικιωμένος, είναι ενεργός, είναι δραστήριος. Είναι δραστήριος απέναντι στους άλλους. Αυτό σημαίνει ότι προσθέτει άλλη μια φάση μεταξύ των γενεών, άλλο ένα στάδιο. Κοίτα την έκθεσή μου. Αναφέρεται σε κοινού τόπους εργασίες που εργάζονται και οι νέοι και οι λιγότερο νέοι. Από τη μία πλευρά έχει ενεργητικότητα, από την άλλη έχει πείρα, από την, ε, έχεις νέες ιδέες από του νέους. Λοιπόν, μπορούμε να είμαστε υγιεί τώρα, ε, κι είμαστε κάπως προχωρημένοι σε ηλικία και αυτό είναι καλό. Έχουμε 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που είναι διαθέσιμο αυτό το σκοπό. Δεν είναι τεράστιο ποσό, αλλά οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στην προσπάθεια. Άρα είναι σημαντικό βήμα, μεγάλο βήμα πρόοδου. Λόγω ελλείψεω χρόνου θα ήθελα να πω κάτι. Στο σημείο 3 ότι ο εθελοντισμό δεν πρέπει να αντικαθιστά την αμοιβόμενη εργασία. Βεβαίω. Ισχύει αυτό. Ότι δεν θα πρέπει αυτοί όμως που κάνουν αυτή την προσπάθεια να, μην, ε, να τους πούμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Ούτε αυτοί που είναι σε μαθητεία και κατάρτιση να χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν ε, θέσεις εργασίας πραγματικές. Λοιπόν, Ρότζερ, μεταδίδεται το πρόγραμμά μας τώρα, η συζήτησή μας και υπάρχουν πολλοί νέοι μπροστά στις οθόνες αυτή τη στιγμή που θα ενθαρρύνονται από αυτά που ακούνε και θα ενθαρρύνονται να κάνουν μια συνεισφορά. Και αυτά που είπες νομίζω ότι τελικά θα είναι Ευχαριστώ κύριο μπουλό και μετά η κυρία Λινκεβιτσιούτα. Κύριο κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Δεν είναι παρόν ο εισήγητης του ΕΛΚ. Εξ ονόματος θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Χάρκιν για τη θαυμάσια εκθεσή του. Δεν μας θέτει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα καταθέσουμε βέβαια κάποιες τροπολογίες. Θέλω να τονίσω ότι ο εθελοντισμός είναι κάτι το πολύ σημαντικό στα πλαίσια μιας καλύτερης κοινωνική ενσωμάτωση εγγράφεται και στη στρατηγική 2020. Επίσης εγγράφεται μέσα στα πλαίσια της ε, καλύτερης γνώσης των καθηκόντων του Ευρωπαίου πολίτη, γιατί νομίζω ότι ο Ευρωπαίος πολίτης μέσα στο έτος 2013 πρέπει να καταλάβει δεν έχει μονάχα δικαιώματα αλλά και καθήκοντα σε σχέση με τους συμπολίτε του και επομένως ο εθελοντισμός είναι ένας ε, τρόπος που βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα το τι σημαίνει να ανήκουμε σε μια κοινότητα και η εθελοντική δραστηριότητα είναι βέβαια τοπική, αλλά μπορεί να υπάρχει και διαμεθοριακού χαρακτήρα εθελοντισμός, ο οποίος αυξάνει το ευρωπαϊκό συνέστημα. Μπορεί κανείς λοιπόν έτσι να μεταλαμπαδεύει εμπειρίες, να δίνει πληροφορίες, να υπάρχει ε, συνεργασία μεταξύ των γενναίων. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Χάρκιν και η ομάδα μας θα ακολουθήσει κατά πάσα πιθανότητα την ίδια γραμμή που ακολουθεί και αυτή με μερικές τροπολογίες μονάχα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία ή ούτε. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ. Τον εισηγητή. Γιατί πρέπει να προωθήσουμε τον εθελοντισμό. Δεν αρκεί να ανακοινώνουμε απλώς ότι κάποιο έτος ονομάζεται έτος εθελοντισμού. Δεν αρκεί αυτό. Διότι αυτή τη στιγμή δεν τα καταλαβαίνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο αυτές τις έννοιες του εθελοντισμού. Μερικές μόλις τώρα αρχίζουν να εφαρμόζουν δραστηριότητες εθελοντισμού, εθελοντιστικές δραστηριότητες και καμιά φορά δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με το θέμα. Αν όμως θέλουμε να πάρουμε απόφαση για την προώθηση του εθελοντισμού αυτό θα ήταν θετικό γιατί θα ενεθάρρυνε και τους γυρεότερους να συμμετάσχουν σε εθελοντιστικές δραστηριότητες. Τους οριμότερους. Τους οριμότερους και τις οριμότερες γιατί αλλιώς μπορεί να βρεθούμε προεκπλήξεων. Τρίτον, αυτό θα ωφελούσε και τους αναπήρους και τις αναπήρους, διότι μπορούν έτσι να εργαστούν από το σπίτι τους εθελοντιστικά. Θα ήθελα να υποστηρίξω τους συναδέλφους που τόνισαν ιδιαίτερα το σημείο 3. Πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά πώς θα αποφύγουμε καταστάσεις όπου ορισμένοι εργοδότες καταχρώνται, εκμεταλλεύονται τον εθελοντισμό για να μειώσουν το κόστος της εργασίας στην επιχείρησή των ή για να αποφύγουν τους φόρους. Η κυρία εισηγήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι συντομότατη γιατί ξέρω ότι μας λείπει ο χρόνος. Καταρχήν, κυρία Ράπτη, συμφωνώ απόλυτα με τα δύο σημεία που θίξατε. Πράγματι όλα αυτά βοηθούν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και δεν πρέπει να υπονομεύσουμε τα υποχρεώσεις του κράτους προνοίας. Για τον Ρότζερ Χάμερ νομίζω ότι είπατε ότι σήμερα γίνατε 68 Εμεί είχαμε ακούσει 60 προηγουμένω, 68. Δεν ξέρω αν είναι τα γενέθλιά σου, αν ναι, χρόνια πολλά. Το τι γίνεται στον έξω κόσμο ε, είναι άλλο θέμα. Δεν ζούμε και σε παράλληλο σύμπαν. Ξέρουμε λίγο πολύ πώ ζει ο κόσμος. Σε ευρωπαϊκό ενωσιακό επίπεδο δεν υπάρχει καμία διευθέτηση για τον εθελοντισμό. Αυτό είναι γεγονός. Μερικοί εθελοντές θέλουν να εργαστούν διαμεθοριακά, μη σε εκπλήσει αυτό. Όσο για τις επιπτώσεις για, πολλούς, για πολλές εθελοντιστικές οργανώσεις, όλα αυτά κάνουν κάποια διαφορά υπέρ τους, το τονίζουν. Για το διαβατήριο ευρωπροσόντων πολλοί νέοι το χρησιμοποιούν και το γράφουν και στα βιογραφικά των. Um, Για την υποστήριξη του CSR τώρα, που λένε είναι κάτι που ωφελεί τις επιχειρήσεις. Όχι, UCSA. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι, περιορίζεται σε δραστηριότητες της μέσης τάξης όπως είπατε, Τόμας. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά που είπες, θα τα συμπεριλάβω. Κύριε Βλόν, αν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε και, και θα το συμπεριλάβω και αυτό, κύριε Μπλινκαβιτσούιτε, για την ενθάρρυνση των οριμοτέρων και των νέων καθώς και των αναπήρων και αυτά τα δέχομαι. Σας ευχαριστώ λοιπόν, άκουσα εξαιρετικές ιδέες και θα φροντίσω να τις συμπεριλάβω στην χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Οπότε έχουμε προθεσμία για τις τροπολογίες μέχρι 31 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι και θα συζητηθούν και θα εξεταστούν στις 29 Φεβρουαρίου. Έχουμε χρόνο. Έχουμε τώρα τις ψηφοφορίες. Έχουμε προσθέσει την προφορική ερώτηση για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Πρώτα απ' όλα θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Κορνέλισεν, που δεν είναι ανάμεσά μας. Πού είναι, δεν τη βλέπω. Έχετε τις κάρτες σας, όλοι. Όλοι. Όλοι. Δεν έχουν πρόβλημα λοιπόν. Παράγραφος 1. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ύψιλον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 3. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Με την παράγραφο 3, νέα παράγραφος που εισάγεται με τροπολογίας 28 του κ. Κοσλόφσκι, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάντα πάνω με την παράγραφο 3, νέα παράγραφος με συμβαστική M λατινικό υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4, συμβαστική Χ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 31 της κυρίας Γιασλοβιέσκα είναι συμβατή, ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται την παράγραφο 4 τροπολογία 32 του κυρίου Πουπάκη καταπίπτει ψηφίζουμε όσον αφορά την παράγραφο 5 την τροπολογία 33 του κυρίου Καμπνόχου, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία, συμβιβαστική ήττα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ξεκινάει ο έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε, πέρας. 21 υπέρ, 18 κατά, μία αποχή. Ε, γκρίνεται. Ε. Μετά την παράγραφο 5, τροπολογία 39 του κ. Καχνόχ κατά αποχές. Έχω την εντύπωση ότι εγκρίνεται, αλλά θα γίνει υπαλήθευση. Λιχτονικός έλεγχος. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 25 υπέρ 15 κατά. Πράγματι εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Συμβαστική, συμβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 καταπίπτει. Ψηφίζουμε τώρα μετά την παράγραφο 6, την 47 σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε πρώτα το κομμάτι commencer par which will, so il y a un problème. Non, ça c'est les mots qui... Ah oui, pardon, pardon. Ok. Alors, donc, nous mettons en voie l'amendement. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 47 σε τμήματα. Όλη την τροπολογία χωρίς το κομμάτι εκείνο το οποίο θα μετακινήσει, which will shift, μέχρι decreasing public deficit. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ προσθήκης του δεύτερου τμήματος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρα να γίνει έλεγχο στο δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι πέρα ψηφοφορία. Δύο ΕΛΚ παραπάνω έχουμε. Κυρία Μπάστο, βγάλτε την κάρτα σα. Εντάξει, εντάξει, τέλο πάντων. 15 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται. Ερχόμαστε τώρα στο τρίτο τμήμα. Όχι, δεν έχει νόημα το τρίτο τμήμα, διότι απορρίφθηκε το δεύτερο. Με την παράγραφο 6 τροπολογία 48 καταπίπτει. Πάμε στην παράγραφο 7 τροπολογία J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Με την παράγραφο 7 τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές έλεγχος νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος Ψηφίσατε όλοι. Τώρα έχουμε τρεις ΕΛΚ παραπάνω. E Δημιουργεί πληθωρισμό, θα το πω στην κυρία Μέρκελ. Δημιουργεί πληθωρισμό το ΕΛΚ. Ακόμα, ακόμα, δεν προσπάθεια. Δύο. Ένα. Ορίστε. Ακόμα ένα παραπάνω. 15 υπέρ, 24 ψήφοι κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 54 του κυρίου Πουπάκη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8 τροπολογία κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για την παράγραφο 7 έχουμε την 57 του κ. Κανόρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 9 έχουμε νέα παράγραφος μέσω συμβιβασμού της Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10, τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 10 συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11, τροπολογία 67 τη κυρία Άρκιν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 12, τροπολογία 68, υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Παράγραφος 13, τροπολογία 69, καταπίπτει, διότι ήδη ψηφίσαμε τη συμβαστική μη, οπότε μετά την παράγραφο 14 έχουμε την τροπολογία 70 του κυρίου Λεγιαρίκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 15 συμβαστική νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 16 τροπολογία συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε μετά την παράγραφο 16 ερχόμαστε στην τροπολογία 77 του κυρίου Καπνόχ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση. Τροπολογία 77 του κυρίου Πουπάκη υπέρ κατά 78 συγγνώμη αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 17 συμβιβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα μετά την παράγραφο 17 στην τροπολογία 83 από την Επιτροπή Γυναικών. Έχει ζητηθεί ξεχωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις εντός των εισαγωγικών. Υπέρ της τροπολογίας 83 χωρίς τις λέξεις των εισαγωγικών κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ της προσθήκης. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 18. Συμβιβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Συμβιβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 19. Τροπολογία 90 του κ. Γιάρη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά την παραγραφό 19 συμβαστική τάφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 19 93 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται την παράγραφο 19 τροπολογία 94 του κυρίου Κοσλόφσκη αυτή καταπίπτει Πάμε στην παράγραφο 20, συμβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 21, δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Μετά την παράγραφο 21, τροπολογία 102 του κυρίου που πάει Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 22, τροπολογία 103 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 22, τροπολογία 104 της κυρίας Γεσλοβιέσκα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται με την παράγραφο 22 τροπολογία 105 Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπότιτλος 4 τροπολογία 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 22 προφορική τροπολογία που σας παρουσιάστηκε χθες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 23, τροπολογία συμβαστική W, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 24, τροπολογία 109 της κυρίας Κορνέλισεν, υπέρ, κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 109 της ηγήτριας. L'inflation Ξανά έχουν πληθωρισμό λόγω ΕΛΚ. Ένας παραπάνω. 2%. 2. Το ΕΛΚ. 21, 18 εγκρίνεται. Καταπίπτει 110, του παράγραφο 24, τροπολογία 111 της ηγητρίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 112 της ηγητρίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 25 τροπολογία 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 25 τροπολογία 114 του Λεγιαρίκ σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα χωρίς τις λέξεις να εκμεταλλευτούν τις συνθήκες εργασίας, τη σκληρότητα των συνδικών εργασίας κλπ. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 114 κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της προσθήκης αυτής της φράσης θα κάνουμε έλεγχο το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 114. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαν όλοι. Πέρας. 22 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα υπέρ της προσθήκης σκληρότης των συνθήκων εργασίας ε, λοιπά Υπέρ κατά αποχές το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 25 τροπολογία 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην ίδια παράγραφο 25 τροπολογία 116 Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 26 τροπολογία 118 συγγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όσον αφορά τις παραθέσεις μετά την 3 τροπολογία 1 υπέρ Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά τη λογική αναφορά 12, τροπολογία 3 της υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 της ηγήτρες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 της κυρίας Κίνγκα Κόλς υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. λογική αναφορά 12, 6, λαμβάνοντα υπόψη το ψήφισμα τη 9η Μαρτίου του 2011 όσον αφορά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την ένταξη των Ρωμά. Ποιο είναι υπέρ αυτή τη τροπολογία 6. Κατά αποχέ εγκρίνεται και αναφορά ε, α, υπέρ, κατά, όσον αφορά τη συμβεστική α, εγκρίνεται. Α, ξέχασα. Μετά τη λογική αναφορά 18 τροπολογία 7, εφόσον και εγώ την υπέβαλα, λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, συμβιβαστική σε λατινικό υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική β υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά τη θεολογική σκέψη σε λατινικό τροπολογία 15 υπέρ, κατά αποχές θα γίνει έλεγχος για την τροπολογία 15 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 15 με 25 απορρίπτεται. Μεγάλη διαφορά. Τροπολογία 16 Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα κάνουμε έλεγχο άρχεται η ψηφοφορία ο ηλεκτρονικός έλεγχος στην τροπολογία 20 ψηφίσατε όλοι πέρας 21 υπέρ 19 κατά εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά Τροπολογία 21, Λεγιάρικ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε το σύνολο της εκθέσεως κ. Κορνέλησεν. Προτείνω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 35 υπέρ. 2 κατά. 2 αποχές. Μπορούμε να συγχαρούμε, πιστεύω, την εισηγήτριά μας. Και πάμε τώρα στη δεύτερη μας ψηφοφορία. Ανακοίνωση της Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την ε, πρόταση προσχώρησης της Σερβίας, αίτηση προσχώρησης της Σερβίας. Έχουμε 8 τροπολογίες εδώ. Τροπολογία 1, Κορνέλσεν, <clears throat> ψήφι Κατά απόχες, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, Κορνέλσεν, υπέρ. Κατά απόχες, δεκτή. Τρία κονέλισεν υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την τρία. Τρία σε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 21-19 εγκρίνεται πράγματι. Τροπολογία 4, Hughes Θέρκας, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 Κονέλσεν υπέρ, κατά δεκτή, 6 Γκένες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 7 κινγκένς κατά αποχές δεκτή, 8 Χιούς θέρκας σε δύο τμήματα. <clears throat> Πρώτο τμήμα, χωρίς τη λέξη όλο, ψήφι υπέρ, κατά Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Α, με συγχωρείτε. Το υπόλοιπο τμήμα της τροπολογίας πρέπει να, να... Μα δεν έχει νόημα αυτό που κάνουμε. Δεν πειράζει τώρα. Τέρα, τι να κάνουμε. Μα έτσι είναι. Δεν έχει νόημα. Ανάποδα τα κάναμε. Η υπόλοιπη τροπολογία υπέρ. Κοτά. Αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα με μεγάλη πλειοψηφία. Συνολική ψηφοφορία. Η προφορική ερώτηση για την ε, εξαίρεση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Πρώτη τροπολογία. Αρκίν Κονέλσεν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία Τη Συρίας Εμού υπέρ <clears throat> κατά αποχές. Τρίτη τροπολογία Τσαμπάορι. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα μπέρες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε μπέρες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου ηλεκτρικά Ψηφίσατε όλοι, όλες, πέρας. 37 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Ωραία λοιπόν. Θέλω να σας υπενθυμίσω τώρα σε όλους τους συντονιστές ότι πρέπει να κινητοποιηθούν αν θέλουμε το θέμα αυτό να εγγραφεί στη μέση διάταξη της Ολομέλες το ταχύτερο δυνατό λόγο και των συζητήσεων στο Συμβούλιο, γιατί δεν είμαστε μέσα στην προθεσμία των τριών εβδομάδων. Αν θέλουμε να γίνει αυτό το Φεβρουάριο, θα πρέπει να κινηθούμε ακαριέως από την πλευρά όλων των πολιτικών ομάδων βασίζομαι στην υποστήριξή σας. Κλείσαμε λοιπόν τις ψ, ψηφοφορίες και περνάμε στο σημείο 25 πρώτο τμήμα της ακροάσεως ημών στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του κανονισμού που διέπει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πρωτού δώσω το λόγο στους κοινωνικούς εταίρους και τις ΜΚΟ που έχουν προσκαλέσει για αυτό το πρώτο τμήμα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μωράν Σαρτιέ που είναι και η συγήτρια. Για να παρουσιάσει την συζήτηση. Σας ευχαριστώ τα μάλα κυρία Πρόεδρε. Σήμερα <clears throat> αντιμετωπίζουμε την τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και φυσικά πρέπει να συζητήσουμε τις γενικές πολιτικές γραμμές της λειτουργίας του Κοινωνικού Ταμείου για τη δημοσιονομική περίοδο μετά το 2013-2014-2020. Θέλω να υπογραμμίσω εξάλλου την σημασία που επέχει για μας όλους και όλες την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Απασχόλησης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης είναι ο κύριος μοχλός που έχουμε <clears throat> στη διάθεσή μας. Mm. Παρακαλώ τους συναδέλφους που έχουν πηγαδάκια να τα μεταφέρουν εκτός της αιθούσης. Παρακαλώ. Κύριε Ορή, και για σας. Ευχαριστώ. Κυρία Μωράν, μπορείτε να συνεχίσετε. Ναι, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και επάγρυπνοι για το θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μετά από το 2003 γιατί, 13, γιατί σε μια εποχή κρίση στο κοινωνικό ταμείο ο κύριο Μοχλό, ο κύριο το εργαλείο που έχουμε για να επιτύχουμε του στόχου για του οποίου έχουμε εργαστεί και έχουμε καθορίσει <clears throat> κατευθυντήρε γραμμέ για την απασχόληση μέχρι το 2020. Υπάρχει μια άρρηκτη σύνδεση μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση τη στρατηγική του 2020, την κινητοποίηση για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό και Ταμείο πρέπει να επιμείνω στον πρώτο στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που είναι φυσικά η επαγγελματική ενσωμάτωση και ένταξη. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι στην πρόταση αυτή υπάρχει ένα τμήμα το οποίο δεν είναι αμεληταίο, 20% δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που αφορά τον αγώνα κατά της ένδυας και επίσης την κοινωνική αλληλεγγύη. 84 εκατομμύρια ευρώ με ένα κανόνα ο πρέπει να τον, οποίο πρέπει να προσέξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το 40% πάντα των πολιτικών συνοχής και μέσα στο Κοινωνικό Ταμείο 20% από τα κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να πάνε για την αλληλεγγύη και το, την καταπολέμηση της ένδυας. Το κοινωνικό ταμείο μπορεί να ενισχύσει όλες τις πολιτικές για την έξοδο από την κρίση που έχουν διατυπωθεί. Τέσσερις είναι οι στόχοι μας, που είναι θεματικού χαρακτήρα και πολύ σημαντικοί. Πρόθεση της απασχόλησης, επαγγελματική κινητικότητα, επενδύσεις στην ανάπτυξη προσόντων και δεξιοτήτων και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και η ενίσχυση των ε, θεσμών και των οργάνων που θα πρέπει να εφαρμόζουν στην πράξη τα προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου. Η πολιτική λοιπόν αυτή εγγράφεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο της ε, εξέλιξης του χώρου απασχόλησης μεταξύ 2014 και 2020 με στόχο να αυξηθεί η, το ποσοστό απασχόλησης, να μειωθούν οι εργασίες χαμηλών δεξιοτήτων και προσόντων, <clears throat> οι ανειδίκευτες επομένως εργασίες, να αυξηθεί το ποσοστό των ε, θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων, συν 15% και φυσικά θα πρέπει να προστατεύσουμε και την, το γενικό πυρήνα των θέσεων εργασίας, το 50% μέσα στις προσπάθειές μας. Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο τα προσόντα και οι θέσεις απασχόλησης θα έχουν σαν κύριο εργαλείο για την επίτευξή του το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ένα δεύτερο λόγο που με ζητά να κινητοποιηθούμε για αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ότι οι πολιτικέ για την έξοδο από την κρίση θα πρέπει να μας επιτρέψουν και να αντιμετωπίσουμε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προβλέπεται ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 27 ότι έχουν εξαφανιστεί από την κρίση και θα πρέπει να ξαναδημιουργηθούν αυτές οι θέσεις εργασίας. Δεν θα είναι φυσικά οι ίδιες θέσεις. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμάσουμε και την κινητικότητα των εργαζομένων και τη δημιουργία νέων προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να δημιουργηθούν εκ νέου θέσει απασχόληση. Ένα δεύτερο φαινόμενο, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, για το οποίο θέλουμε επίση να κινητοποιηθούμε από την Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Θεμάτων, είναι το γεγονό ότι οδοτούνται πολύ. Το baby boom, η μεγάλη γενιά του μεταπολέμου και εκεί θα πρέπει να ανανεώσουμε τις γνώσεις και τα προσόντα και αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο γεγονότα μιλάμε <clears throat> για περίπου 60 εκατομμύρια θέσεων εργασίας που θα πρέπει μέχρι το 2020 να ανανεωθούν. Βλέπουμε λοιπόν ποια η σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σχετικά. Μεταξύ τώρα των θεμάτων για τα οποία έχουμε κάνει ειδικέ ακροάσεις με τους καλεσμένους μας στους σημερινούς και στα οποία είναι σημαντικά στα οποία θέματα σημαντική συνεισφορά τους είναι τα εξής. Καταρχήν, το θέμα των ρητρών επιλεξιμότητος και ιδιαίτερα η ρήτρα επιλεξιμότητος που έχει να κάνει με την μακροοικονομική κατάσταση διότι υπάρχει αυτή η αίτηση να εξαρτηθεί η πορεία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου από την καλή διαχείριση στο εσωτερικό των κρατών μερών. Μετά από την ανακοίνωση του ε, Επιτρόπου Αντόρ για το θέμα αυτό, εγώ ετάχθην σαφώς κατά μια τέτοια ρήξας επιλεξιμότητας. Εγώ υποστηρίζω τον χρυσού κανόνα. Υποστηρίζω την καλή διαχείριση στα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν η χρήση των Ταμείων Συνοχής και Χωροταξίας, αλλά, αλλά στο Κοινωνικό Ταμείο είναι διαφορετικά τα θέματα, μας ενδιαφέρει η ένταξη των εργαζομένων, δεν μπορούμε να φανταστούμε να υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ μακροοικονομικής εξέλιξης και κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, μια πολύ σημαντική συζήτηση για την οποία εμεί θα πρέπει να εκφέρουμε μία σαφή θέση και θα μας βοηθήσουν σίγουρα οι εταίροι μας. Το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να αναφέρω είναι η απλοποίηση των κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Χρειαζόμαστε σχέδια. Γνωρίζουμε ότι στην πράξη δεν χρησιμοποιείται πάντα πλήρω το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην κινητοποίηση αυτών των πόρων. Τρίτον, θέλουμε να έχουμε ε, μετρήσιμα στοιχεία για τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είναι σημαντικό ο ρόλος του Κοινωνικού Ταμείου για τη δυναμική τη απασχόληση. θα πρέπει όμω να τύχει καταμέτρηση και να συμφωνήσουμε σε σχέση με τα κριτήρια και τους δείκτες που θα μας επιτρέπουν, όχι να λέμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά να δούμε με αντικειμενικό τρόπο κατά πόσο είναι επιτυχής οι πολιτικές μας. Εν συντομία λοιπόν τα λέω αυτά κυρία Πρόεδρε, έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα και έχουμε να πούμε και περισσότερα σε σχέση με την ενσωμάτωση των κοινωνικών εταίρων, σε σχέση με τη χρήση του κοινωνικού ταμείου Ήδη, ήδη μέσα σε μια ομάδα εργασία μας με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα κάναμε πολλές ακροάσεις για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας γιατί είναι πολυεπίπεδη η ανάγκη να εμπλέξουμε τους κοινωνικούς εταίρους ιδιαίτερα σε επίπεδο επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ λέει κυρία Μπερές. Πριν ή δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας, θέλω να προτείνω να μην ασχοληθούμε με τη μακροοικονομική εξάρτηση στην ακρόαση και μόνο, γιατί υπάρχει μια ευρεία συνένεση στην Επιτροπή μας και η οποία επιδεινούται, αν θέλετε, από το γεγονός ότι αν δείτε τι έχει προκύψει από το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ για τις διεθνείς συμφωνίες, για τη διακυβερνητική μάλλον συμφωνία, υπάρχει τώρα δυνατότητα κυρώσεων με ένα ποσοστό του ΑΕΠ που εγγράφεται στην διακυβερνητική συνθήκη. Επομένως, <clears throat> ήδη έχει δημιουργηθεί μια ρύθμιση αυτού του είδους. Δεν θέλω λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί υπάρχουν πολλαπλέ άλλε πτυχέ οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και δεν θα πρέπει να παίξουμε κρυφτούλη σε σχέση με άλλα σημαντικά στοιχεία. Θα δώσω πρώτα τον λόγο. Για 10 λεπτά στο, στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων η κυρία Κλοντ Κενακ Γκάου που είναι σύμβουλος της Συνομοσπονδίας. 10 λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εκ νέου ευχαριστώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας των συνδικάτων που μας καλέσατε σε αυτή την ακρόαση και που την διοργανώσατε επί ενός θέματος που είναι θεμελιώδου σημασίας για την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Συνδικάτων, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αν αληθεύει ότι είμαστε τακτική επαφή επί του θέματος με την ομάδα την κοινοβουλευτική ε, είναι ξεκάθαρο πρέπει να, ξε... υπογραμμίσουμε κάποια ε, θέματα στα πλαίσια συνεδριάσεων των Επιτροπή Απασχόλησης. Εν πρώτης, δεν θα επικεντρώσουμε όλη τη συζήτηση ευτυχώς σε αυτή τη μακροοικονομική εξάρτηση. Ε, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, όπως ήδη υπόθηκε, ότι είναι απαράδεκτο, τουλάχιστον για μας, να τίθενται όροι μακροοικονομικοί που είναι εις βάρος μέσω των κυρώσεων προσωρινά και μόνιμα την κακή διαχείριση την πολιτική που ασκείται κακή σε κεντρικό επίπεδο, ομοσπονδιακό κλπ. Και αυτό είναι κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες για τις περιφέρειες, την τοπική αυτοδιοίκηση και για τους πολίτες. Και αυτό δημιουργεί ευρωσκεπτικισμό στον πληθυσμό των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωσκεπτικισμό που αυξάνεται μετά την οικονομική κρίση και κυρίως μετά τα μέτρα λιτότητας που έχουν ληφθεί και θεσπιστεί από τις Βρυξέλλες όπως παρουσιάζεται διότι δεν εξηγείται σωστά από τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε προτάσεις για να δημιουργηθούν κάποιοι κοινωνικοί όροι και εξάρτηση. Δεν μιλάμε για την οικονομική διακυβέρνηση και όλα τα σχετικά προγράμματα που θίξατε. Δεν μιλάμε για την κοινωνική πτυχή, για την κοινωνική διακυβέρνηση, αυτό που ζητούμε. Θέλουμε μια κοινωνική προσέγγιση χωρίς εξαρτήσεις, δηλαδή την εφαρμογή και το σεβασμό των πλήρη της αρχής της εταιρική σχέσεως στα πλαίσια όλων των διευθυντικών ταμείων. Τι σημαίνει αυτό. Την εφαρμογή και το σεβασμό των οδηγιών των ευρωπαϊκών νόμων στους κοινωνικούς τομείς. Όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, την απόσπαση των εργαζομένων, που είναι επίκαιρο θέμα, πολύ επίκαιρο. Την ισότητα των φύλων και να μην πω τόσες λεπτομέρειες. Καταλάβατε που το πάω. Δεύτερον, όσον αφορά το γενικό κανονισμό. Ανησυχούμε διότι στο Γενικό Κανονισμό των Διεθνωτικών Ταμείων δεν αναφέρεται καθόλου πλέον η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Εμφανίζεται στη συνθήκη, ευτυχώς, στη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά πλέον δεν εμφανίζεται καθόλου στην πρόταση του κανονισμού για τα διεθνωτικά ταμεία και θα πρέπει, είναι απαραίτητο, να επανενταχθεί, να συμπεριληφθεί. Παρόλο που σε συναντήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα εξηγούν ότι πρόκειται περί γραφειοκρατικού σφάλματο, τεχνικού, τιούτου κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά. Ξέρουμε ποια ρεύματα κινούνται σε κάποιες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. Για να επανέλθουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αυτό κάθε αυτό, και στα μέτρα που θίξατε σε σχέση με τα αποτελέσματα. Δηλαδή, προσέγγιση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για την αποδοχή των προγραμμάτων και για την αξιολόγηση της εφαρμογής τους, υλοποίησεώς τους. Έχουμε μεγάλες επιφυλάξεις και αμφιβολίες. Και ας είναι ξεκάθαρο ότι τα μία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, είναι τα μία που χρηματοδοτούν τα τσέπη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι σαφές τι πρέπει να κάνουμε, όπως και όλα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, αλλά να συνδέουμε την έγκριση ενός προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικά Ταμείο με τα αποτελέσματα, για να γίνει αυτό χρειάζονται σωστοί δείκτες, συγκεκριμένοι. Διότι είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε τα αποτελέσματα αν κατασκευάζεται ε, ένας δρόμος ή μια γέφυρα. Στα εγγένεια βλέπω τα αποτελέσματα από το να δει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αφορά την απασχόληση που βρέθηκαν ή διατηρούνται μετά από μια κατάρτιση για τους νέους ή για τους ανθρώπους που είναι μακριά από τον τόπο εργασίας και που γίνεται προσπάθεια επανένταξης και για νέους με λίγα ή καθόλου προσόντα. Χρειάζονται λοιπόν σαφέστατε δείκτες. Το επεξεργαζόμαστε το θέμα που συμπεριλαμβάνονται εν μέρη αυτή στο παράρτημα της προτάσεως του κανονισμού. Όσον αφορά την θεματική συγκέντρωση, όπως τη λέει στην ορολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τέσσερις προτεραιότητες. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτές τις προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα η απασχόληση και εν μέρη κινητικότητα. Αυτό μπορούμε να το ξανακουβεντιάσουμε εν συνεχεία. Μετά έχουμε δεύτερον ένταξη ε, αν θα πετύχουμε τους στόχους του 2020, να μειώσουμε τουλάχιστον σε 20 εκατομμύρια αυτούς που είναι φτωχοί, που ξέρουμε ότι έχουν αυξηθεί παραπάνω μετά τη λήψη της από το Συμβούλιο λόγω οικονομικής κρίσης, λόγω συνεπιών της οικονομικής κρίσης. Τρίτος στόχος, κατάρτιση. Ανθρώπινη πόρη. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κυρίως στον αφορά τους νέους. Τέταρτον, ενίσχυση της διοίκησης και της αποτεσματικότητας των διαφορών διοικήσεων, και όσον αφορά την κατάρτιση. Πολλοί υπάλληλοι δεν έχουν υποστεί την κατάρτιση, δεν είναι αρκετά ενήμεροι όσον αφορά τους νόμους, τις δυνατότητες που υπάρχουν. Και υπάρχει έλλειψη. Ε, πρέπει να μειωθεί, να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία, να υπάρξει απλούστευση για την κινητικότητα φερειπίν των εργαζομένων. Ε, των ερευνητών, των σπουδαστών. Συμφωνούμε ότι το ότι καθαρίζουμε 20% των ποσών των, κοινωνικών ταμείων να μπουν για την καταπολέμηση της ένδυας για την κοινωνική ένταξη, θα θέλαμε εξίσου να θέσουμε στο 40% τα ποσά των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Ταμείων που θα αφιερώνονται για τις πολιτικές απασχόλησης για την ενίσχυση των εν λόγω πολιτικών και την προσπάθεια για την ένταξη. Με όσα αυτά συνεπάγονται, χωρίς να περιοριζόμαστε προφανώς τις κατευθύνες γραμμές για την απασχόληση. Κάποιες που απομένουν στις ολοκληρωμένες κατευθύνσεις που ψηφίστηκαν και ψηφίζονται τακτικά από το Συμβούλιο. Να επιμείνουμε εκ νέου για να αναφέρουμε εκ νέου μια ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόληση. Όχι μόνο επί χάρτου, αλλά και επί χάρτου. Δεν ξέρω αν το διαπιστώσατε στα έγγραφα που μα δίνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναφέρεται πλέον. Ευρωπαϊκή στρατηγική λοιπόν ήταν απασχόληση που πραγματική ήταν και εκτιμένο μετά την κινητοποίηση και τη διεκδίκηση της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας των συνδικάτων και των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν. Άλλο θέμα σημαντικό η νέα έννοια των περιφερειών σε μεταβατική φάση δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αυτό σαν έννοια. Είδαμε εξηγήσει που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν αρκούν. Δεν είμαστε εκ των προτέρων κατά της νέας αυτής ενίας, αλλά θα θέλαμε για, τα, για τις περιφέρειες σύγκλησης να υπάρχουν και άλλα κριτήρια πέρα από το περίφημο 75% το ΑΕΠ το μέσο όρο, να υπάρχουν κριτήρια που αφορούν το ποσοστό ανεργίας της περιφέρειας, ε, συμμετοχή στα σχολεία κλπ. Πάρα πολλές παράμετροι και δείκτες πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, για να καθορίζεται το επίπεδο ανάπτυξης, ας είμαι θετική, ανάπτυξης των περιφερειών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να υπάρξει ανοιχτή προσέγγιση προς περιφέρειες. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες, οι πιο αδύναμες περιφέρειες να μην βρίσκονται σε ισχυρή θέση. Να λάβουμε υπόψη επίσης ότι τώρα, επί του παρόντος τώρα με την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε, δεν ξέρουμε αν οι σημερινές πλούσιες ε, περιφέρειες θα γίνουν φτωχές αύριο. Ελπίζουμε ότι πλέον ε, φτωχές ε, περιφέρειες να είναι λιγότερο φτωχές στο μέλλον. Η οικονομική κατάσταση μας οδηγεί σε σύνεση, πρέπει να είμαστε συνετοί. Και ο κανονισμός που συζητούμε, που θα ισχύει μετά το 2013, ελπίζουμε ότι τότε όταν θα ισχύσει θα έχουμε βγει από την οικονομική κρίση. Βλέποντας όμως τα στοιχεία που έχουν διάθεσή μας καθημερινά, τα πρόσφατα στοιχεία, επιτρέψτε μας να έχουμε κάποιες αμφιβολίες ή τουλάχιστον να πάρουμε όλα τα μέτρα τόσο ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Άλλο στοιχείο που αφορά το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ναι θα ολοκληρώσω τώρα, για μας είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα αντίθετα από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό το Ταμείο να μην είναι ανοιχτό για ενισχύσεις ε, προς τους γεωργούς που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Υπάρχουν άλλοι πόροι γι' αυτό. Υπάρχει η κοινή αγροτική πολιτική, ο πυλώνας ο δεύτερος που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και που θα πρέπει να χρησιμοποιείται ακόμα περισσότερο για αυτές τις πολιτικές της απασχόλησης ή καταπολέμησης της ανεργίας ή επανένταξης. Και δεύτερον, επιμένουμε επί το εξή. Οι αρχές και οι στόχοι του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που, σε, που αναδιορθώνονται να προσθεθούν στους στόχους τους, της προλήψεως που βρίσκουμε στα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία με τα προβλεπόμενα κονδύλια. Και τέλος, κάτι που δεν είναι ασήμαντο, η εταιρική σχέση, είμαστε ικανοποιημένοι που υπάρχει αυτή η πρόταση διοντολογικού κώδικα. Κατά κάποιο τρόπο ήταν διεκδίκησή μας και ήταν και στη γνωμοδότηση της οικονομική Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Δεν αρκεί όμως, δεν είναι δεδομένο και όσον αφορά το περιεχόμενο είναι σημαντικό να υπάρχει ευρωπαϊκός ορισμός της εταιρικής σχέσης για να μην ακολουθούνται εθνικές πρακτικές σε κάποιες χώρες. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν πρακτικές εσωτερικές πάνω σε αυτό και γίνεται ό,τι τους κατέβει, χωρίς να λέω τώρα λεπτομέρειες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σαφής ορισμός του ρόλου και των λειτουργιών κάθε εταίρου. Και εν πάση περιπτώσει ο κοινωνικός διάλογος ε, είναι αποκλειστικό προνόμιο των κοινωνικών εταίρων. Ό,τι σχετίζεται με την πολιτική απασχόληση, ορισμός, η διαχείριση της απασχόλησης είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων και πάνω σε αυτό νομίζω ότι μπορώ να πω ήδη ότι συμφωνούμε απόλυτα εμείς οι κοινωνικοί εταίροι. Και τέλος, ζητήσαμε και κλείνω ότι η διαβούλευση ε, δεν διοργανώνεται σωστά, ούτε επαρκώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αυτή η προσήκηση. Έγραφαμε στον πρόεδρο τη Επιτροπή Μπαρόσο και στον επίτροπο, τον υπεύθυνο για τον προπολογισμό και τον επίτροπο Αντόρ και Χάν, ούτω ώστε να φροντίσουν, ούτω ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν ζητήσει σωστά, όχι μόνο όσον αφορά τι προτάσει που αφορούν τις δημοσιονομικέ προοπτικέ, αλλά όσον αφορά όλο το πακέτο που αφορά την ε, πολιτική κοινωνική, οικονομική και εδαφική ε, συνοχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και Συγγνώμη, δεν είχα δει το χρόνο ε, δεν θέλω να κάνω διακρίσεις εναντίον των επόμενων ομιλητών, απλώς δεν είχα παρακολουθήσει το ρολόι. Για το ΠΕΜ, κυρία για 10 λεφτά και πάλι. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Απασχόληση για το γεγονό <clears throat> ότι μα προσκαλέσατε να δώσουμε τη γνώμη μα για το νέο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που προτάθηκε από την Κομισιόν και είναι τώρα να συζητήσει στο Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο. Για, για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει και εμπλοκή των ε, ε, υπευθύνων των εμπλεκομένων από την πραγματική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν λοιπόν να δώσουν τη γνώμη τους για το μέλλον. Τα διαδοτικά ταμεία και ιδιαίτερα το κοινωνικό ταμείο είναι σημαντικά και απαράγραπτα εργαλεία για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση τώρα και θα είναι και στο χρονικό διάστημα 2014-2020. Έρχομαι τώρα στα σημεία τα οποία Μα έχετε ζητήσει να διεξέλθουμε και είναι σε δύο τμήματα η παρουσίασή μου. Πρώτα υπογραμμίζω την θετική αξιολόγηση, τα σημεία που είναι θετικά και το δεύτερο, δεύτερο τμήμα αφορά τα πιο αρνητικά σημεία. Σε επίπεδο θετικό ξέρουμε ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο δέσμευση κονδυλίων στα διαδοτικά ταμεία και στο κοινωνικό ταμείο για να επιτευχθούν οι στόχοι των προτεραιοτήτων της Ευρώπης 2020. Χαιρετίζουμε και το νέο <clears throat> πακέτο κανονισμών για τα θέματα αυτά. Πιστεύουμε ότι η προσέγγιση αυτή... Συγγνώμη, πήδησα μια σελίδα και χάσα τις πίσω μου σελίδες. <clears throat> Χαιρετίζουμε λοιπόν το νέο πακέτο κανονισμών μεταξύ των οποίων και ο τρέχον κανονισμός. Τρίτον, Χαιρόμαστε που υπάρχει ένας πολιτι... ένας... Ε, ένα κονδύλιο του προπολογισμού για ανταγωνιστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα τον υπογραμμίζουμε τη σημασία της ευθυγράμμισης με τους στόχους της Ευρώπης 2020, καλύτερη ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, καλύτερη απασχόληση, διαβίου μάθηση και κοινωνική συμπερίληψη. Ω εκ τούτου, συμφωνούμε απόλυτα στους εξής 7 χώρους που είναι κάτι που πάντα διεκδικήσαμε. Την αρχή της συγκέντρωσης. Μία συγκέντρωση σε προτεραιότητες. Η απασχόληση όμως και ο αγώνας κατά της ανεργίας θα πρέπει να είναι η πρώτη, η πρώτη προτεραιότητα, ιδίως για τους νέους, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για αυτούς. Δεύτερον, χαιρόμαστε για τη νέα ε, προσέγγιση που υπάρχει στην αρχή στην αρχή της Κομισιόν και επίσης για τις νέες μορφές διακυβέρνησης και το γεγονός ότι υπάρχει ένα άρθρο για όλα τα ταμεία. Τρίτον, για τη συνεργασία που θα υπάρξει μεταξύ κυβερνήσεων για τα πολιετή προγράμματα. Χαιρετίζουμε επίσης τους στόχους της Κομισιόν να εξασφαλίσει ε, διοικητική απλοποίηση, ιδίω στην e την πρωτοβουλία e-commit, για να γίνεται ηλεκτρονικά δέσμευση των κονδυλίων. <clears throat> Έκτον, υποστηρίζουμε και τα προγράμματα που έχουν σαν στόχο να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους παρά τις, ε, την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ δημοσίων αρχών και διαχειριστών για να πετύχουμε να εφαρμοστεί αυτή η νέα προσέγγιση, κάτι που δεν είναι εύκολο. Και επίσης ζητούμε να αναπτυχθεί περισσότερο η ικανότητα των κοινωνικών εταίρων ώστε να μπορέσουν επαρκώς να διαδραματίσουν το ρόλο που τους αρμόζει ως κέρι παίκτες στο <clears throat> εγχείρημα αυτό. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο κομμάτι της παρέμβασής μου, τα πιο προβληματικά στοιχεία για την εταιρική σχέση. Θα θέλαμε να είναι πιο σαφής ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα, να είναι, υπάρχει ανταγνώρισή τους, ιδίως για τους θεματικούς στόχους, την κάλυψη της απασχόλησης και της παιδείας και επίσης για τη διαβίου ε, εκπαίδευση και τις δεξιότητες για την καλή διακυβέρνηση και τη σωστή εφαρμογή της εταιρική σχέση θα θέλαμε να έχουμε και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων τουλάχιστον σε διαβουλευτικό επίπεδο στον κώδικα συμπεριφοράς και το κοινό πλαίσιο πολιτικής. Και επίσης θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για τους στόχους μας να τονιστούμε ότι πρέπει να υπάρχει μνήα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου <clears throat> σε όλους τους κανονισμούς όπως γίνεται τώρα. Προτεραιότητες θέλουμε να δώσουμε μια σαφή μνήμα στον θεματικό στόχο 3 της επαγγελματικής κατάρτισης και αυτό είναι και ο θεματικός στόχος 10 στο γενικό κανονισμό. Επίσης, μια νέα πρωτοβουλία επενδύσεων στις μαθητείες. Είναι πολύ σημαντική η μαθητεία για να προωθηθεί η απασχόληση. Και εν τέλει θα θέλαμε να έχουμε να αναφέρονται οι τα η μετακίνηση μεταξύ των, ε, επιχειρήσεων και επίσης η δημιουργία επιχειρήσεων και το επιχειρήν. Συμπεράσματα είμαστε εν γέννη ικανοποιημένοι με την πρόταση της Κομισιόν και τώρα εναπόκειται στο Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο να βελτιώσουν το κείμενο αυτό και παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία και τέλος Εμείς θα σταθμίσουμε τη θέση μας σε σχέση με το πακέτο των οργανισμών και θα τη δώσουμε στη διάθεσή σας εν καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο το, για, για τις επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, ο κύριος David Ancien, Ancien, συγγνώμη, έχετε το λόγο για ένα δεκάλεπτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνεται να εκφράσουμε απόψη μας για το, για, το μέλλον των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Ταμείων και να γίνει ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συζητάμε σημαντικό θέμα για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, κυρίως τώρα τους καιρούς ε, δημοσιονομικών περιορισμών. Γίνονται περικοπές στους προπολογισμού και οι βασικές ε, γίνονται περικοπές στις βασικές υπηρεσίες, οι επενδύσει ε, αναβάλλονται, να μην πω ότι κινούνται σε όλη την Ευρώπη, ακούμε ότι γίνονται σοβαρέ περικοπέ στην παιδεία, στην περίθαλψη, την υγειονομική, στι υποδομέ. Αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη όλο και περισσότερο βραχυπρόθεσμες πολιτικές και αυτό είναι ανησυχητικό για το μέλλον. Τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία και εν γέννη η πολιτική της ε, συνοχής είναι τα βασικά εργαλεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βασικός κλάδος οικονομικός και πολιτικός που έχει μακροπρόθεσμα αντίκτυπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά προσεκτικά, κυρίως εν ώψη της επερχόμενης διαβούλευσης που θα γίνει για το στρατηγικό πλαίσιο. Εγώ εκπροσωπώ τους εργοδότες της επιχειρήσεις που παρέχουν ε, ε, δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη ή κοινοφελείς υπηρεσίες. Ανάλογα με τους όσους χρησιμοποιείτε, μπορείτε να καλέσετε. Αυτές χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία. Σχόλια για τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία. Πρώτον, ευπρόσδεκτη διασύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Ταμείων με τη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 για βιώσιμη και ενταξιακή ανάπτυξη. Η Ευρώπη έχει στρατηγική για τα επόμενα χρόνια και πρέπει να την εφαρμόσουμε. Έχει σαφή στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαφή στόχους, φιλόδοξους στόχους απασχολησιμότητα 75%, μείωση κάτω από 10% και φεύγουν τα σχολεία και 40% τουλάχιστον των νέων να έχουν κάποιο πτυχίο υψηλού επίπεδου. Και υπάρχει συσχετισμός μεταξύ όλων των, όλων των κοινωνικών ταμείων. Άρα και το, εάν υπάρχει μεγαλύτερη συνδιασύνδεση, υπάρχει και μεγαλύτερο φαινόμενο μόχλευσης. Πρέπει να πλουστευτούν οι διοικητικέ διαδικασίε. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται σωστή ισορροπία μεταξύ υποβολή εκθέσεων και ελέγχου και να μπορούν όμω και πιο ελεύθερα τα στελέχη να αποφασίζουν για τις δραστηριότητέ του. Θέλουμε αποδοτικότερη διαχείριση. Συχνά επιχειρήσει δεν έχουν χρόνο να ζητήσουν καν και να διεκδικήσουν και να υποβάλουν αιτήσει για τη χρηματοδότηση που χρειάζονται. Καμιά φορά η αρχική επένδυση είναι πολύ μεγάλη για τις επιχειρήσεις. Σημαντικό να γίνει απλούστευση. Καλό είναι να χρησιμοποιηθούν κατά αποκοπήν ποσά, κυρίως. Και να δούμε και από άλλα προγράμματα τι γίνεται. Όσον αφορά την αξιολόγηση, και να δούμε πώς θα γίνεται η πραγματική αποτίμηση των ε, εφαρμογή των προγραμμάτων. Πρέπει να είναι σαφές και να αναφέρεται το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι δημόσιες ε, υπηρεσίες που παρέχονται. Όχι μόνο σαν ιδέα, όχι να φαίνεται σαν πνεύμα στη, στα κείμενα σημασία που έχουν τις υπηρεσίες. Χρειάζεται και στήριξη οικονομική που θα ανταποκρίνονται και στις ανάγκες και στους στόχους. Στην παρούσα κατάσταση, την οικονομική, τα ευρωπαϊκά κοινωνικά ταμεία πρέπει να είναι σημαντικό στρατηγικό και οικονομικό εργαλείο, να διαθέτουν πόρους για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις για τις επενδύσεις και τις προτεραιότητες αυτών. Να πω κάποια πράγματα. Θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις για την καταπολέμηση των αποτελεσμάτων της κρίσεως. Επενδύσεις σε δεξιότητες και σε εκπαίδευση. δεν υπάρχει αντιστοιχία σωστή μεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών. Υπάρχει μεγάλη ενεργία, αλλά υπάρχει και έλλειψη δεξιοτήτων και ταλέντων. Έγινε κάποια έρευνα πρόσφατα που το έδειξε αυτό. Μπορεί να καθυστερήσουν στρατηγικές πρωτοβουλίες λόγω ελλείψεως δεξιοτήτων. Περίπου 15% των επενδύσεων των ενεργειακών χάνονται λόγω ελλείψεως του κατάλληλου εργατικού δυναμικού. Στην Ευρώπη, παρά την κρίση, υπάρχουν πολλές καινές θέσεις, διότι δεν υπάρχουν ε, επαρκείς δεξιότητες. Και το πρόβλημα είδαμε να αυξάνεται το 2010 και το 2011. Στι δημόσιε υπηρεσίε είναι ακόμα σημαντικό το φαινόμενο. Γιατί χρειαζόμαστε ιδιαίτερε δεξιότητες και γνώσεις. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη γύρανση του εργατικού δυναμικού. Και στον τομέα μας είναι μεγαλύτερος ο μεσόρος ηλικίας από τις άλλες τομείς. Και πολλοί από αυτού που του εργαζόμενου θα βγουν στη σύνταξη την επόμενη δεκαετία. Οι δημογραφικέ αλλαγέ είναι σημαντικέ για το μέλλον, πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γίνονται προβολέ από τη Eurostat. Ο μέσο όρο θα παει 40-48 μέχρι το 2016. Και θα μειώνει το αριθμό των νέων. Και θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Αύξηση του κόστου των κοινωνικών συστημάτων αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και επίσης η μεταβιβασιμότητα των προσόντων. Οι ουσιώδεις υπηρεσίες πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι συνεχώς αυξάνονται λόγω των κοινωνικών αλλαγών. Για όλους αυτούς τους λόγους αλλά και άλλους θέλουμε και εμείς να συμβάλλουμε στη συζήτηση με το Κοινοβούλιο για το μέλλον αυτού του σημαντικοτάτου θέματος. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο για τους μήκη όμικρον στον κύριο Κονιρόιτερ. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας μιλήσουμε εδώ πέρα. Δεν είναι εδώ κοινότοπο το πρόγραμμα που συζητάμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ουσιώδες για την αντιμετώπιση της κρίσης. Γιατί άμα δεν βρούμε τη λύση τότε θα καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι οι όροι με τους οποίους ε, εφαρμόζεται, αλλά το, η ίδια η χρήση των κοντιλίων, η κατάχρηση η κακή χρήση. Πρέπει να δούμε πρώτα πού βρίσκονται οι ανάγκες. Πού είναι η αναποτελεσματική διαχείριση και διοίκηση. Ποιες είναι οι ανάγκες για την εκπαίδευση, για την απόκτηση προσόντων κλπ. Όλοι συμφωνούμε νομίζω ότι πρέπει να στοχεύει το κοινωνικό ταμείο εκείνους που πραγματικά το χρειάζονται. Όπως είπε και στην αρχή της ε, παρουσίασής της η Πρόεδρος. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε την προσθετικότητα λοιπόν. Είναι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν έχει νόημα να τιμωρήσουμε αυτούς που χρειάζονται βοήθεια και τις χώρες που πρέπει να αναπτυχθούν και να πούμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κοινωνικό ταμείο. Μείο. Καλό είναι επίσης θα ήταν στα πλαίσια του κοινωνικού ταμείου να αναφέρουμε δύο βασικά σημεία. Ένα το είπαν οι προηγούμενοι. Δεν μιλάμε πια για την στατική της απασχόλησης. Ενώ οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η Ένωση δεν ασχολείται ούτε με την απασχόληση ούτε με τα κοινωνικά. Αν θέλουμε να συνδεθούμε με τους πολίτες πρέπει να δούμε να καταλάβουμε ότι το κοινωνικό ταμείο έχει και αυτό μια πολιτική πτυχή. Επίσης η στρατηγική του 20 έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τη δημόσια συζήτηση και πρέπει να επανέλθει διότι η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται σε αυτήν. Εμείς οι κοινωνικές μήκοι όμικρον είμαστε υπέρ της στρατηγικής του 2020. Θέλουμε όμως να υπάρξει ολόκληρη ανάπτυξη, όχι τμήματική. Προτείναμε λοιπόν και εμεί, μία δική μας εξάμετρο, όχι τη δική σας το six μία άλλη. Προτείνουμε λοιπόν ένα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να στοχεύει κυρίως κοινωνικούς στόχους. Νομίζω εδώ συμφωνείτε οι περισσότεροι και να απλοποιηθεί, να δει ποια είναι οι προτεραιότητες της κοινωνικής καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανέχειας. Επίσης να τονίσουμε ιδιαίτερα θέματα ισότητας των δύο φύλων και ίσης μεταχείρισης διότι γνωρίζουμε ότι σε περιόδους κρίσης το θέμα της άνησης μεταχείρισης αυξάνεται το πρόβλημα. Δεύτερον, η γενική χρηματοδότηση. Είμαστε υπέρ και καμιά φορά η Κομισιόν θεωρεί ότι οι μήκοι όμικρον δεν είναι διαχειρίσιμες. Όχι, όχι, είναι, είναι. Θα θέλαμε απλώς το 25% των ταμείων συνοχής να αναφέρεται στην γενική διευθέτηση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει για το πολυετές πλαίσιο, αλλά αυτή η ρήτρα του 25% είναι κάτι στο οποίο επιμένουμε έπειτα. Είμαστε υπέρ της χρησιμοποίησης του 20% για από το Κοινωνικό Ταμείο για την καταπολέμηση της ανέχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν πρέπει να σκεφτείτε καμία μείωση περαιτέρω. Τέταρτον, το θέμα των εταιρικών σχέσεων. Ναι, με τους φίλους μας, τους κοινωνικούς εταίρους, ακούμε συνεχώς ότι το θέμα της απασχόλησης είναι θέμα κοινωνικού διαλόγου. Αλλά εκείνοι που δεν παίρνουν μέρος στο κοινωνικό διάλογο γιατί δεν έχουν προσόντα ή είναι εκτός της αγοράς εργασιάς ή δεν βρίσκουν δουλειά που να αποκρίνεται στα προσόντα τους, πρέπει και αυτοί να επανέλθουν στον διάλογο, να βρουν μία έναν προσανατολισμό. και κατά κάποιον τρόπο να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας στις οργανώσεις μας. Εδώ και 25 χρόνια ασχολούμαστε με αυτό. και για μας αυτό προέχει η καταπολέμηση του αποκλεισμού. Αυτό δεν έρχεται σε αντίφαση με τη συνεννόηση των κοινωνικών εταίρων, είναι συμπληρωματικό. συμπληρωματικό. όχι μόνο αυτές οι συνεργασίες αλλά και η χρηματοδότηση των μήκη όμικρων. Σήμερα οι οργανώσεις αυτές που ασχολούνται με την επαγγελματική κατάρτιση δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση ή αυτό διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα και δεν έχουν πρόσβαση γιατί σε μερικές χώρες όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά και αλλού, για πολιτικούς λόγους οι κοινωνικές μήκη ε, όμικρον αποκλείονται από την πρόσβαση σε τέτοια κονδύλια. Αν θέλουμε να κάνουμε πράγματι κάτι, όπως είπαν και οι εργοδότε, πρέπει να συνδυάσουμε τις ανάγκες τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Υπάρχει ανάγκη να λάβουμε υπόψη μας και όσους αποκλείονται ή κοντεύουν να αποκλειστούν από αυτήν. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό οι μικρές ιδιαίτερα οργανώσεις μέσω της απλοποίησης που ζήτησε η κυρία Μωρέν Σατνέ να μην καταλήξει αυτή να αποκλείσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των κοινωνικών μήκη όμικρων. Πόσο έχω ακόμα, τρία λεπτά, τέσσερα λεπτά. Και ξέρω ότι θα τα να συζητήσετε αυτά, αλλά για μας αυτές είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να έχει το κοινωνικό ταμείο. Τι θα στοχεύσουμε ιδιαίτερα, τη νεολαία που δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή και όσους είναι άνω των 55 γιατί η Ένωση θέλει να τους ενεργοποιήσει και αυτούς. Σήμερα τι γίνεται, άμα κανείς είναι 50, 52 ή 55 τον διώχνουνε ή δεν βρίσκει δουλειά. Πρέπει λοιπόν το κοινωνικό ταμείο όχι μόνο να είναι καλύτερα στοχευμένο για τους νέους αλλά και για τους πιο ηλικιωμένους και για τους μετανάστες και μετανάστριες τι θα γίνει. έχουν ίσως χαρτιά ή δεν έχουν χαρτιά αλλά είναι εδώ και δουλεύουν εδώ. Επίσης θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο και για τα προσόντα και δεν εννοούμε μόνο τις βιομηχανικές θέσεις εργασίας αλλά και τη φροντίδα Δεν το λέω πρώτη φορά, αλλά μας αρέσουν οι προτάσεις που ακούγονται και οι τροπολογίες για τη βελτίωση των θεμάτων της φροντίδος. Σας ευχαριστώ ακόμη μία φορά που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι όντως πολύ ωφέλιμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταίο προσκεκλημένος για το πρώτο τμήμα αυτής της ακροάσης και εξ του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Αένδιας, η κυρία Σιαν Τζόνς, η οποία είναι πολιτική συντονίστρια στο δίκτυο αυτό. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση εν συντομία για το δίκτυο κατά της ένδυας. Είμαστε ένα ανεξάρτητο δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων κατά της ε, ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχουμε 13, 30 μάλλον, yeah. Ναι. πλατφόρμες σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, 23 από τις οποίες είναι από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτούς που δεν ξέρουν τα λέω αυτά. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας με σαφήνεια ότι για μας οι προτάσει τη Κομισιόν σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι μέσα από τα πιο θετικά και απτά αποτελέσματα του στόχου, των στόχων της Ευρώπης 2020. Όλη μας η προσπάθεια και η άσκηση πίεσης για την καταπολέμηση της έχουν <clears throat> ευδοκιμήσει. Μέσα στο προτάσεις της Κομισιόν εμείς χαιρετίζουμε το γεγονός ότι υπάρχουν δύο σαφείς χώροι, η ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της ε, ένδειας, δηλαδή το ότι προσδιορίζεται 20% των κονδυλίων για τη μείωση της ένδειας Και το δεύτερο στοιχείο που υποστηρίζουμε είναι η αρχή της εταιρικότητας και η αρχή της προσέγγισης εκ των κάτω. Να υποστηρίξουμε τοπικές πρωτοβουλίες, να υποστηρίξουμε την ε, απλοποίηση και συστήματα που να είναι πιο φιλικά στις ΜΚΟ. Θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους στόχους και θα επανέλθω σε λίγο σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους. Ένα τέταρτο στο μέσο θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι δεν μπορεί μόνο του το κοινωνικό ταμείο να λύσει το πρόβλημα της ένδυας. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους διαφορετικούς πόρους. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχουμε μια ρήτρα για mainstreaming των κοινωνικών θεμάτων και έναν τρόπο να καταμετρούμε την πρόοδο προς τους στόχους αυτούς για την καταπολέμηση της για το θέμα της εξάρτησης. Χαιρόμαστε που και η Επιτροπή σας έχει απορρίψει διαρρήδην την ιδέα αυτή της μακροοικονομικής εξάρτησης. Θέλω να εστιάσω τώρα ιδιαίτερα στο γιατί, στο τι μπορεί να κάνει μάλλον το Κοινωνικό Ταμείο για να εξασφαλίσει αποτελεσματική λειτουργία του στόχου για τη μείωση της ένδυας. Είναι απαραίτητο να κινηθούμε με βάση το 20% το οποίο είναι υπό πίεση και κίνδυνο. Θέλω να τονίσω λοιπόν γιατί είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το 20% για την αντιμετώπιση της ένδυας. Πρώτα απ' όλα η Κομισιόν έχει αναγνωρίσει ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω βελτίωση. Η στρατηγική έρευνα λέει ότι η πρόοδος για την επίτευξη του στόχου της μείωσης ένδυας είναι βραδής. Βραδία η πρόοδος και δεν έχει καλύψει όλους τους στόχους. Δεύτερον, μόνο 12% αυτή τη στιγμή του κοινωνικού ταμείου χρησιμοποιείται για την κοινωνική συμπερίληψη. Είναι χαμηλό ποσοστό. Και το πιο σημαντικό η κοινωνική, κοινωνικός αποκλεισμός και η ένδια αυξάνονται λόγω της κρίσης και τώρα λόγω των μέτρων λιτότητας. Η νέα έκθεση της Κομισιόν η οποία παρακολουθεί τον κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης και η οποία θα αντιμετωπιστεί στο Συμβούλιο Κορυφής του Φεβρουάριου λέει ότι πάνω από 2 εκατομμύρια ατόμων είναι σε κίνδυνο ε, να πέσουν στο χώρο της ένδυας. Όχι μόνο αυτό, αυξάνει και το βάθος της ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 340.000 άτομα ακόμα αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα υλικής αποστέρησης. Και αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου μονάχα. Υπήρξε αύξηση στους εργαζόμενους φτωχούς κατά 8,5% στα 8,5% από 8%. Αυτό είναι το 1 τέταρτο των εργαζόμενων, των ατόμων σε ε, ηλική εργασίας που είναι ενδέης. Η εργασία δεν τους βγάζει από τη φτώχεια. Χρειάζονται νέοι πόροι. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα απασχόλησης αλλά και επέκεινα της απασχόλησης. Πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Αυτό σημαίνει πρέπει να έχουμε περισσότερε επενδύσει για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Επίση, ο προσδιορισμό του 20% εξασφαλίζει και την εδαφική <clears throat> συνοχή. Είναι απαραίτητο για να έχουμε μια ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των χωρών και αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκεται υποκίνδυνο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα εξασφαλίσουν ότι αυτό το 20% παραμένει στην κύρια προτεραιότητα της καταπολέμησης της ένδυας. Κάτι ακόμα που θέλω να πω για την επιστημιστική βοήθεια. Προς το παρόν η πρόταση είναι ότι το σύστημα επιστημιστικής βοήθειας θα είναι μέσα στο 20%. Δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς υποστηρίζουμε την επιστημιστική βοήθεια, αλλά αυτό δεν είναι στρατηγική αντιμετώπισης της ε, ένδυας. Είναι μια πυροσβεστική ενέργεια η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει την τρομερή κατάσταση που υπάρχει τώρα. Δεν πρέπει αυτό να αντικαταστήσει τα μέτρα πολίμησης της ε, ένδυας. Τονίζουμε πρέπει να είναι μια πρόσθετη γραμμή του προπολογισμού και πάντα χρηματοδοτείται εκτός των διαχρονικών ταμείων. Πρέπει να είναι χωριστό λοιπόν κονδύλι. Ο δεύτερος χώρος που θέλω να τονίσω είναι η ανάγκη να κάνουμε πιο σαφείς τις προτεραιότητε και τους θεματικού στόχους για την καταπολέμηση τη ένδυα. Χαιρόμαστε για την εστίαση στην απασχόληση, αλλά αυτό σημαίνει για μας μόνιμη και ε, ποιότητα και απασχόληση ποιότητας. Όπως είδαμε, δεν φτάνει η απασχόληση για να βγάλει τους ανθρώπους από την ένδια. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στην απασχόληση, όχι μόνο το να διατηρήσουμε αυτούς που εργάζονται και μια πανάκια, μια γενική προσέγγιση δεν αρκεί για όλους. Πρέπει να θέσουμε στοχευμένους ε, στόχους κατά περίπτωση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ομάδες οι οποίες έχουν πολλαπλά προβλήματα και μειονεκτήματα. Η ενεργή συμπερίληψη είναι μία από τις θετικές προτεραιότητες, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Έχει τρεις πυλώνες αυτή τη στιγμή. Επαρκή υποστήριξη στα εισοδήματα, προσωπική υποστήριξη για, έργο, εργασία ποιότητας και ποιοτικές υπηρεσίες. Έχουμε τρεις πυλώνες λοιπόν και δεν πρέπει να βασιστούμε μονάχα στην ενεργή ε, απασχόληση και δεν πρέπει να τα μπλέξουμε αυτά με την επιλεξιμότητα. Σας λέω και πάλι η απασχόληση είναι κέρια, αλλά θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη με την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, ιδίω υπηρεσίες. Ένας τέταρτος τομέας είναι η προσέγγιση με το στόχο της Ευρώπης 2020 και ευθυγράμμιση με τους στόχους αυτούς σίγουρα το υποστηρίζουμε γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τους στόχους της μείωσης της ένδυας. Θα πρέπει να δοθεί όμως ίση ε, σημασία στο στόχο της φτώχειας και με τους άλλου στόχους γιατί φοβόμαστε ότι αυτή τη στιγμή η έμφαση είναι, έμφαση περισσότερο σε άλλους στόχους. Επίσης, <clears throat> για να επιτευχθεί αυτό χρειαζόμαστε ένα σύστημα κοινωνικής αξιολόγησης που θα εκτιμήσει τον βαθμό στον οποίο το κοινωνικό ταμείο επιτυχάνει του στόχους αυτούς. Χρειαζόμαστε να έχουμε όχι μονάχα μετρήσιμους δείκτες, αλλά και η πρόοδος για την αντιμετώπιση της κοινωνικής, ε, του κοινωνικού αποκλεισμού, ήπιοι λοιπόν δείκτες για όλα αυτά τα θέματα και καλύτερη σύνδεση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού. Το ξεχνάμε αυτό, υπάρχει μια κοινωνική μέθοδο συντονισμού με στόχους, με μια σειρά δείκτων για τα αποτελέσματα και όλα αυτά θα συνδέονται με τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης, τις εθνικές κοινωνικές εκθέσεις. Με μια καλύτερη σύνδεση θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αλλά και πάλι πρέπει να τονίσω ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή της μακροοικονομικής εξάρτησης θα θέσει ένα αμφιβόλο όλα αυτά τα στοιχεία και θα δώσει μόνο έμφαση στη συμμόρφωση με την μακροοικονομική παγίωση. Αυτό είναι διπλή ε, τιμωρία. Όχι μόνο για όλη την κοινωνία, αλλά και για τις πιο αδύνατες ομάδες. Τέλος, είναι σημαντική η μνήμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αναγνωρίζει η πρόταση ότι οι ΜΚΟ έχουν την απαραίτητη εμπειρία για να εργάζονται με τροτές ομάδες του πληθυσμού και ομάδες ατόμων που, που είναι αποκλεισμένοι από την κοινωνία. Και είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε την επανεζωμάτωση όλων αυτών των ανθρώπων και τη συμμετοχή του στην κοινωνία. Προ το παρόν έχουμε πολλή εμπειρία με άτομα τα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πόρου του κοινωνικού ταμείου. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο όμω κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η συμμετοχή των εταίρων σε όλα τα πλαίσια, σε όλα τα επίπεδα τη ε, διαδικασία, στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση είναι απαραίτητο. Πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε την ιδέα της εταιρικής σχέσης, να τονίσουμε την τεχνική αρρωγή που είναι απαραίτητη για να βοηθήσει τις μικρές ΜΚΟ να επωφεληθούν από τα ταμεία αυτά και πρέπει να κάνουμε προσβάσιμα τα συστήματα αυτά ώστε να μπορούν να έχουν συνολική χρηματοδότηση. <clears throat> και πρέπει να δημιουργήσουμε και το σύστημα δημιουργίας ικανοτήτων πέραν των κρατών μελών και για άλλους φορείς οι οποίοι έχουν προτεραιότητα. Σε επίπεδο Απλοποίηση Εμείς χαιρετίζουμε τις προτάσεις αυτές και τονίζουμε ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν περισσότερο μηχανισμοί φιλικοί προς τους ΜΚΟ. Κατά αποκοπήν ποσά, απλοποιημένες διαδικασίες και ένα ακόμα στοιχείο που είναι ελλείπων κρίκος είναι οι καθυστερημένες πληρωμές. Δημιουργεί μεγάλη δυσκολία για τις ΜΚΟ γιατί αναγκάζονται να χρεώνονται ένα τελευταίο θέμα επίσης είναι το θέμα της διεθνικής συνεργασία, το οποίο αναφέραμε προηγουμένως. Χαιρετίζουμε αυτές τις προτάσεις, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να επιτρέψουμε να υπάρχουν και διεθνικά και διαμεθοριακά σχέδια τα οποία φέρονται σε πέρα από ΜΚΟ. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη λοιπόν υποστήριξη σε όλα αυτά τα δίκτυα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ήταν πληρέστατη η παρουσίαση μου λέγουν ότι δεν μπόρεσαν να παραστεί η Business Europe, δεν υπήρξαν εκπρόσωποι που να μπορέσουν να παραστούν και συμβάλλουν στην συζήτηση ανεξαρτήτως της θελήσεώς μας συμβαίνει αυτό. Θα ακολουθήσουμε τη σειρά με την οποία δήλωσαν ενδιαφέρον να μιλήσουν οι συνάδελφοι. Ο κ. Τόμας Μαν πρώτος και μετά ακολουθεί ο κ. Νταρντέν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής διότι μπορούμε να περάσουμε τα... Πάμε στα 80-84 ε, δισεκατομμύρια. Αυξάνονται τα χρήματα, δεν θέλουμε να σπαταληθούν, να χρησιμοποιηθούν σωστά θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στις δράσεις μας να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα. Εξεπλάγει, διότι αναφέρθηκε ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλαμε κοινό output, κοινή εκροή με τους δείκτες που έχουμε εισάγει. Από παλιά τους είχαμε δημιουργήσει. Ε, είδαμε τι λειτουργήσε σε κάποιες χώρες, κάναμε απολογισμό, είδαμε τι πήγαινε καλά και τι δεν πήγαινε καλά και χρειαστήκαμε ένα εργαλείο που να μας επιτρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάθαμε από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι σε κάποια κράτη-μέλη η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν λειτουργήσε καλά. Γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει να πούμε ότι ένα μέρος των χρημάτων του Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει διατίθεται για την αύξηση του δυναμικού για να βοηθούνται οι κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις των καταναλωτών για να συμμετέχουν καλύτερα στις διεργασίες. Είναι πολύ σημαντικό να το φροντίσουμε αυτό. Να αναπτυχθούν δυνατότητες, να δημιουργηθεί δυναμικό, να υπάρχουν δυνατότητες κατάρτισης, ευαισθητοποίησης, να γίνει κατανοητό πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι. Οι δεμοί θα κινούμεθα εν κενό. Είναι πολύ σημαντικό. Όλα τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου ζητούν πάντα την ενίσχυση των κοινωνικών εταίρων είναι συνήθεια αυτή, είναι πρακτική που ακολουθούμε και είναι απαραίτητο να γίνει αυτό και στα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι εσείς μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτό. Έχω μία ερώτηση προς την Ελίζαμπετ. Έχουμε ενδιαφέρουσα έννοια που αναφέρθηκε και θέλουμε να υποστηρίξουμε την κοινωνική καινοτομία. Είναι πολύ σημαντικό. Περί τίνος πρόκειται όμως, τι είναι κοινωνική καινοτομία, πού τη βλέπουμε, τι καινοτόμο υπάρχει θα ήθελα τα διάφορα κοινωνικά μέτρα που ε, εφαρμόζονται να έχουν αποτελέσματα. Αλλά να λέμε έτσι γενικά ότι τα μέτρα είναι ε, καινοτόμα είναι υπερβολικό. Θέλουμε απλούστευση. Να δούμε πώς λειτουργεί αυτή. Να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Όλοι προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Και εμείς οι ευρωβουλευτές ε, δεχόμαστε πολλέ καταγγελίε και διαμαρτυρίε από τον κόσμο που μα λέει ότι δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Πρέπει να πετύχουμε αποτελέσματα. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έχει προτεραιότητα αυτό. Ε, Κλείνοντα, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθούμε επί 4-5 βασικών προτεραιοτήτων να τι εφαρμόσουμε πραγματικά. Να μην έχουμε πολλέ προτεραιότητε. Να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε λιγότερε. Και αν γίνει αυτό θα είναι καλή δουλειά. Χτες είχαμε την κυρία Μωρά και εδώ ε, οι Γάλλοι είναι πολύ παρόντες στη συζήτηση των θεμάτων αυτό και είναι πολύ καλό. Ο κύριος Νταρντέν και μετά η κυρία Γιασοβιέτκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους προσκεκλημένους και προκεκλημένες μας είναι βασικό το θέμα που συζητάμε για την κρίση που αντιμετωπίζουμε και που φαίνεται ότι δυστυχώς θα συνεχίσει. Σημερίζομαι πολλά από αυτά που άκουσα. Ιδιαίτερα το 20% για την καταπολέμηση της ανέχειας στο Ταμείο. Αυτό συνεχίζει και την έκθεσή μας για την καταπολέμηση, την περσινή μας έκθεση για την καταπολέμηση της ανέχειας. Χαίρομαι επίσης για την έννοια της μεταβατικής περιφέρειας ή περιοχής. Πρέπει όσο δυνατόν περισσότεροι πολίτες να υποφεληθούν από αυτά τα ταμεία. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για να μπορέσουμε να κρίνουμε την αξία των μέτρων και σχεδίων γιατί η αποτελεσματική χρήση είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Εδώ χρειαζόμαστε ό,τι προτάσεις μας κάνουν, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα διαθέσιμα ταμεία Ζητάμε μεν όλο και περισσότερα και αυξάνονται όντως, αλλά πρέπει να ξέρουμε και ποια είναι η καλύτερη δυνατή χρήση τους. Επίσης, ο καλύτερος συντονισμός των ταμείων. Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πρέπει να διατηρήσει την ιδιαιτερότητά του όπως και όλα τα άλλα ταμεία. Και τέλος, καλό θα ήταν νομίζω να ενδυναμωθούν οι αποστολές και τα κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου ιδιαίτερα για την διατροφιμική βοήθεια γιατί επεκτείνοντας, παρατείνοντας τις αποστολές καταλήγουμε τελικά να μειώνουμε τα κονδύλια. Επομένως, αυτή η ιδέα του 40% για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι κάτι που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Έπειτα, αν και η πρόεδρος δεν θέλει να επιμείνουμε σε αυτό, το θέμα της άρνησης της προσθετικότητας είναι κάτι που και αυτό πρέπει να συζητηθεί. Ευχαριστώ. Γεια Σλοβιέτκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ συχνά επικρίνουμε την αποτελεσματικότητα με την οποία χρησιμοποιεί το Κοινωνικό Ταμείο. Χθε η κυρία Μωρέα οργάνωσε πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες και που μας έδειξαν ποια ήταν η διαφορά μεταξύ δεξιοτήτων, προσόντων και απαιτήσεων ε, της αγοράς εργασίας. Ερώτηση. Μπορούν να γίνουν, να εφαρμοστούν καινοτόμες δράσεις ούτως ώστε να προσαρμαστούν οι δεξιότητε και τα προγράμματα κατάσταση που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στι ανάγκε αγορά εργασία. Στην περιοχή μου οργανώσαμε ένα πρόγραμμα με, Γερμανούς, με τους Γερμανούς εταίρους μας και μία φορά κάθε τρει μήνες οι επιχειρηματίες της περιοχής μας έδιναν πληροφορίες. Οι πληροφορίε αφορούσαν τι ανάγκε του, όσον αφορά τους εργαζομένους, τι προσόντα χρειαζόταν τι είδο εργαζομένους θα απέλυαν. Αυτό το πρόγραμμα συλλογή πληροφοριών από του εργοδότε δυστυχώ σταμάτησε. Πέρασαν έκτοτε 14 χρόνια. Έχουμε αρκετές πληροφορίες η λέξη για να πετυχαίνουμε καλύτερη κατάρτιση. Το χρειαζόμαστε αυτό. Αν είχε συνεχίσει το πρόγραμμα θα είχαμε κάποια στοιχεία ε, που θα μας επέτρεπαν να αντλήσουμε διδάγματα για το μέλλον. Να ξέρουμε τι θα χρειαζόμαστε. Έχετε πληροφορίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εν ώψη των νέων προοπτικών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για να χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι πόροι και να βοηθήσουμε εκείνους που βρίσκουν προβλήματα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η κυρία Σρέτερ τώρα έχει το λόγο και μετά η κυρία Κίνγκεν Κούντς. Σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε. Θα ήθελα να υποβάλω ένα αίτημα. Να στείλετε γραπτό στις ε, πανεβάσεις σας. Προσπάθησα να σημειώσω αυτά που λέγατε όταν μιλάγατε, αλλά μου ξέφυγαν πολλά. Ε, έπιασα όμως κάποιες πολύ καλές συγκεκριμένες προτάσεις που ήθελα να τις μελετήσω και να τις λάβω υπόψη για να τροπήσουμε τον κανονισμό. Λοιπόν, παρακαλώ τις προτάσεις σας αν μπορούσατε να τις υποβάλλετε γραπτός. Ε, ένα άλλο έχω να πω. Ότι αναφέρθηκαν κάποια πράγματα ε, τα οποία παίζουν ρόλο μεγαλύτερο στον γενικότερο κανονισμό από ότι στον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν για μένα να μας στείλετε γραπτός στις προτάσεις σας και σε αυτές να αναφέρετε τι θα θέλετε να αλλάξει στο γενικό κανονισμό, στον κανονισμό πλαίσιο όσον αφορά την απασχόληση, κοινωνική ένταξη, καταπολέμηση της ανέχειας κλπ. Διότι υπάρχουν θέματα αφορούν χρηματοδότηση, χρηματοδότηση, κανόνες για τα οικονομικά ζητήματα. Όλα αυτά αντιμετωπίζονται στον κανονισμό πλαίσιο και άλλα στον ειδικό κανονισμό. Αληθεύει ότι υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη, πλειοψηφία, που θέλουν ε, να μην γίνεται αυτή η αναφορά και πιστεύω ότι πάντα η Επιτροπή Απασχόλησης, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω στο Κοινοβούλιο, που υποστηρίζει ε, καθορισμό κάποιων ορίων. Πρέπει να τα υπενθυμίσουμε λοιπόν αυτά. Αυτό που με εξέπληξε είναι ότι σε καμία από τις παρεμβάσεις σας δεν τονίζεται παρκώς οι διαφορές που υπάρχουν στο άρθρο 6 όσον αφορά την εταιρική σχέση έχουμε καλή έννοια τις εταιρικέ σχέσεις για κάποιες χώρες αναφέρεται αλλά δεν μιλήσαμε γενικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι η εταιρική σχέση αυτό είναι σημαντικό κατά την άποψή μου ίσως θα μπορούσατε να ξαναμιλήσετε πάνω σε αυτό για την επιστημιστική βοήθεια τι θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό όταν ζητάμε να δημιουργηθεί κονδύλι να... συμπληρωματικό, εγώ θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ουτοπία. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά χρήματα για τα άλλα εργαλεία. Και γι' αυτό είναι ουτοπικό να κάνουμε αυτό που λέτε. Υπάρχουν απ' την άλλη έξι κράτη-μέλη που είναι βασικοί συνεισφορείς για τη χρηματοδότηση από 1η πρώτου 2014 αυτά τα χρήματα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εν ώψη του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Λοιπόν, εάν ακολουθήσουμε τον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είχαμε ένα πλεονέκτημα. Θα ήταν καλύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. θα μπορούσαν να συνδυαστούν η επιστημιστική βοήθεια με άλλα μέτρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Καλό θα ήταν λοιπόν, καλή ιδέα να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αυτές οι ενισχύσεις. Τέλος. Εξεπλάγιν, διότι δεν αναφερθήκατε εκτενώς το θέμα της συγκέντρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αναφέρθηκε έτσι ακροθυγώς αυτό το πρόβλημα και θα πρέπει να εξετάσουμε το σημείο 4 που αναφέρονται τέσσερις θεμελιώδεις προτεραιότητες του άρθρου 9 του κανονισμού, πλαισίου, του γενικού κανονισμού. Αυτό αρκεί. Πρέπει να περάσουμε 4 σε 5 προτεραιότητες από 4 σε 6, να μην έχουμε καμία. Δεν ελοχεύει ο κίνδυνος μιας διάχυση ε, ε, διασπάθηση των πόλων αρκεί να λέμε τέσσερις προτεραιότητες εκ των οποίων η μία πρέπει να εφαρμοστεί ε, πιο προσεκτικά. Θέλω συγκεκριμένες δηλώσεις όταν μιλάτε και όχι γενικόλογα, διότι αυτό θα πρέπει να, συγκεκριμένα πράγματα θα πρέπει να γράψουμε και να συμπεριλάβουμε στον κανονισμό. Η ε, κυρία Κίνκεν Κούντς και μετά η κυρία Χάρκεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο το ότι γίνεται αυτή η ακρόση. Και η επόμενη είναι σημαντική. That... Ακούγοντας τα σχόλιά σας έχω την εντύπωση ότι είναι σημαντική αυτή η συνεργασία που ίσως θα έχουμε. Συνεργασία εκείνων που επεξεργάζονται ως εισηγητές και ως εισηγητές επί του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Κοινοβούλιο και εκείνων από εσά που γνωρίζουν πολύ καλά το πώς εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα και έχουν συστάσεις να μας κάνουν. Όπως είπε η Εύα Σρέντερ, νομίζω θα ήταν πολύ χρήσιμο για μας αν μας στέλνατε και σε μένα προσωπικά ακόμα συστάσεις, γραπτός, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε συστάσεις, προτάσεις, σκέψεις σας για να τις χρησιμοποιήσουμε. Μιλάμε για τον κανονισμό ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι σημαντικό να εναρμονίσουμε αυτό το κανονισμό με τον κανονισμό πλαίσιο. και οι συνάδελφοι της Επιτροπής Ρέτζι και οι άλλοι συνάδελφοι που εξετάζουν τα θέματα καινοτομία και κοινωνικών αλλαγών και σχετικό κανονισμό να υπάρχει επαφή με όλους αυτούς για να εργαστούμε όλοι μαζί και να εναρμονίσουμε τους κανονισμούς. Να πω και κάτι άλλο. Το εδαφικό σύμφωνο και την έννοια της εταιρικής σχέσεως και την αρχή, τη σχετική. Αυτή η αρχή είναι πολύ σημαντική και θα είναι σημαντικότητα η εφαρμογή τη και η παρακολούθηση τη εφαρμογή τη από πλευρά Ευρωπαϊκή Επίτροπή, Διότι μιλώντα για εταιρική σχέση, όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάμε παρά να εφαρμόζεται και να βλέπουμε να υλοποιείται επιτόπου αυτή. Σε τοπικό επίπεδο, νομίζω ότι χρειάζεται επεξεργασία. Επεξεργασία των λεπτομεριών τη εταιρική σχέση, τη ενία εταιρική σχέση και των εδαφικών συμφώνων, περιφερειακών συμφώνων. Πώ να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, κυβερνητικέ οργανώσει κλπ. Από τη μια βλέπω ότι χρειαζόμαστε σωστή αποκέντρωση της εφαρμογής για να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Το είπατε κι εσείς. Η χρήση του ταμείου πρέπει να είναι αποτελεσματικότερη. Ταυτόχρονα, απ' την άλλη, χρειαζόμαστε στεναρότερο έλεγχο πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ενώση αφορά του στόχου, τι εθνικέ στρατηγικέ. Θα θέλαμε να εφαρμόζονται εθνικέ στρατηγικέ σύμφωνα με κανόνε για να πετύχουμε τους στόχους του 2020. Και τα επιχειρησιακά προγράμματα να παρακολουθούνται κατά πώς εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων. Είναι σημαντικότατο να ακολουθήσουμε τα ποσοστά που αναφέρονται, 25% του Ταμείου Συνοχής για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 20% να ακολουθούν τα ποσοστά που αναφέρονται για τα, και για τα προγράμματα προτεραιοτήτων. Το Συμβούλιο, από ό,τι γνωρίζω, και κάποια κράτη-μέλη δεν είναι ικανοποιημένα πραγματικά με τα ποσοστά αυτά, τα δεσμευτικά. Θα ήταν σημαντικότατο να υποστηρίξετε εσείς, όλοι οι οργανισμοί σας, αυτή την προσέγγιση. Το σχέδιο πρότασης δεν είναι καλή και η ομάδα εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ήταν ένα πολύ καλό πλαίσιο για στενέ επαφέ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τη σύνταξη τη πρόταση. Στόχο μα τώρα να παραμείνουν τα θετικά στοιχεία απλούστευση των κανόνων, ούτω ώστε το κοινωνικό ταμείο να είναι προσβάσιμο για μικρού φορεί, να έχουν άμεση επαφή με τις ομάδες της κοινωνίας που πραγματικά χρειάζονται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και η εναρμόνιση του Ταμείου είναι πολύ σημαντική για να συσταθούν περίπλοκα προγράμματα για τις τοπικές κοινότητες. Μέχρι τώρα υπάρχουν ε, ε, προγράμματα με υποπρογράμματα και όχι συνάθρηση περίπλοκων προγραμμάτων. Μπορούμε να υποστηριχθούμε. Στείλτε μας ε, προτάσεις. Πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζονται και οι κανόνες στον κανονισμό πλαίσιο. Και πρέπει να εξετάσουμε και τι γίνεται και στον κανονισμό για κοινωνική αλλαγή. Αρκίν, αν θέλει κανείς άλλος να μου το πει, ε. Μπάστος. Κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών και ομιλητριών. Χάρκιν. Ευχαριστώ όλους και όλες. Μιλήσατε για μεταβατικές περιφέρειες. Πρέπει εδώ να είμαστε προσεκτικοί και ευέλικτοι. Συμφωνώ ότι μέχρι τώρα λέει να πάρει το έτο, τα έτη 7 με 9 ως έτη αναφοράς αλλά σε πολλές περιφέρειες μόλις τώρα φαίνονται στους αριθμούς τους τα αποτελέσματα και μπορεί να καταλήξουμε τελικά να βάλουμε περιφέρειες ως μεταβατικές που δεν είναι και να μην βάλουμε άλλες που είναι λόγω των αποτελεσμάτων της κρίσεως. Δεν ξέρω τι ευελιξία θα μπορούσαμε να προβλέψουμε, αλλά ευελιξία πάντως. Είναι πολύ ωραία αυτή η εναλλακτική πρόταση εξαμέτρου σε εναλλαγή με τη δική μας. Συμφωνώ με την Κίνγκα ότι δεν αρκεί μια γενικόλογη νομοθεσία, χρειάζονται και οι λεπτομέρειες. Να αναλύσουμε πώς λειτουργεί η αρχή της εταιρικότητας, σε ποιες χώρες μέλη, από το 4 και μετά υπήρξε το έγγραφο με τίτλο «Η αυταπάτη της η αυταπάτη της συμπερίληψης και πρέπει να το ξαναδούμε αυτό για να είναι όλα σίγουρα τα στοιχεία. Πολλές από τις λεγόμενες πρωτοβουλίες που στηρίζονται σε κοινότητες βασίζονται σε θελοντές, αλλά τι ακριβώς χρηματοδότηση έχουν. Άλλοι. Many of them are overstretched, they're borrowing from banks, etc. Α, μίλησαν για καθυστερήσεις πληρωμών. Είναι σοβαρό πρόβλημα για τους μήκη αυτό. Και έχουν εμποδιστεί πολλές δραστηριότητες τους από τις καθυστερήσεις αυτές. όταν εγκρίνεται μια δαπάνη πρέπει να πληρώνεται γρήγορα. Άλλοι μίλησαν για ολοκληρωμένη προσέγγιση των συμπεριλήψεων. Αν έχετε καμιά ιδέα να μου την πείτε. Τέλος. Άλλος μίλησε για κακό συνδυασμό προσόντων. Αυτό το εξέτασε και το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και κατ' εκείνους, πολλοί εργαζόμενοι έχουν υπερβολικά προσόντα και άλλοι πολύ λίγα. Και δεν έχουν συνδυαστεί οι δύο αυτές κατηγορίες. Πρέπει να τα θέσουμε όλα αυτά σε περιφερειακή βάση και ατομική ακόμα. Τι έχετε να μας πείτε και γι' αυτό. η κυρία Μπαστός. Θέλετε να λάβετε το λόγο τώρα κυρία εισηγήτρια ή μετά το τέλος συζήτησης. Ναι, ναι, όχι αμέσως. Η κυρία Μπαστός και αμέσως θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες και μετά στην κυρία Μωρά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είχα ήδη εκδηλώσει τη θέλησή μου να λάβω μέρος σε αυτή τη συζήτηση που είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση και θέλω να συγχαρώ την κυρία Μωρέν Σαρτιέ και όλους τους προσκεκλημένους της που παίξαν σημαντικό ρόλο στην εξέταση αυτού του θέματος και μας βοήθησαν να καταλάβουμε όλες τις πτυχές αυτού του κανονισμού, του, των νέων κανονισμών. Οι στόχοι που έχουν καθοριστεί είναι πραγματικά οι μεγάλοι στόχοι που θέλουμε εμείς να επιτύχουμε με το ευρωπαϊκό κοινωνικό επίπεδο. Ο στόχος μας είναι να διοχετεύσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα κονδύλια ώστε να προωθήσουμε την ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας και να αντιμετωπίσουμε το γενικό επίπεδο ανεργίας που είναι πολύ ψηλό και που είναι μια πραγματικά δραματική απόρρεια της οικονομικής και της κοινωνικής κρίσης που ζούμε στις χώρες μέλη μας. Η, κοινωνική, η, η επαγγελματική κοινοτικότητα, η επένδυση στα κοινωνικά θέματα και αυτά προτεραιότητες πρέπει να λάβουμε υπόψη με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η επένδυση για καλύτερα προσόντα είναι πάλι ένας τρόπος να βελτιώσουμε την αγορά εργασίας μας και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί με καλύτερους ανθρώπινους πόρους στην συνολική <clears throat> οικονομία που απαιτεί όλο και μεγαλύτερο δυναμισμό και επομένως όλο και καλύτερη κατάρτιση σε επίπεδο εφαρμογών. Ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη η σωστή εφαρμογή επιτόπου και αυτή μπορεί να αλλάξει τα πράγματα οι τοπικές αρχές και οι εθνικές αρχές βέβαια πρέπει να έχουν σαφείς στόχους και προσωπικό το οποίο είναι καλά εξοπλισμένο και εκπαιδευμένο για να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Η σωστή παροχή συμβουλών σε τοπικό επίπεδο και η χρήση των πόρων που βρίσκονται κοντά στους πολίτες και που είναι απαραίτητη για τη σωστή αξιοποίηση αυτών των πόρων είναι αποφασιστικού χαρακτήρα. Επίσης, λόγω <clears throat> της ε, μεγάλης ανεργίας και την έλλειψη πόρων, η δική μου χώρα έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τα θέματα αυτά. Τέλος, δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι απορρίπτουμε διαρρήδην όλη την αρχή της ε, εξάρτησης από τη μικροοικονομική ε, και εξάλλου θέλουμε να εξασφαλίσουμε και την απλοποίηση στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και επειδή έρχομαι από ένα κράτος μέλος το οποίο βρίσκεται κάτω από το βάρος των μέτρων λιτότητος ότι τα μέτρα αυτά του κοινωνικού ταμείου θα πρέπει να βοηθήσουν να ξεπεράσουμε όχι μόνο την ανεργία αλλά και τις ανισομέρειες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέτοντας σε κίνδυνο ορισμένες περιοχές που είναι αυτές που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο της σύγκλησης και επομένως εκεί θα πρέπει να δοθεί έμφαση από τα ταμεία. Τέλος, η ενσωμάτωση των κοινωνικών εταίρων, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορέσει να υπάρξει μια ισοδίκαια εφαρμογή των ε, πόρων των ταμείων αυτών. Πρέπει να υπάρξει πλήρης δέσμευση και συμπερίληψή τους από την αρχή μέχρι την εφαρμογή των σχεδίων και με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσουμε ότι γίνεται πραγματικά η παροχή των πόρων αυτών στους πραγματικούς αποδέκτες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις πριν το κάνω αυτό, να καθησυχάσω τους δύο που είναι για το επόμενο σημείο τη διάταξη, κύριο Άντερσεν και κύριο Μεζιέρ. Θα συμπεριλάβουμε τα σημεία τους για τα οποία είναι ανάμεσά μας με λίγη καθυστέρηση. Μην ανησυχούν. Μην ανησυχούν. Έχουμε κερδίσει λίγο χρόνο βάσει με την αλλαγή που κάναμε χθε και θα έχουν στη θέση του το χρόνο προβλεπόταν τα κουρασή του χωρί προβλήματα. Αλλά θα θέλαμε να συζητήσουμε, να τελειώσουμε σωστά την πρώτη συζήτηση. Mm, mm, mm. που εμπίπτει πλήρω η συζήτηση αυτή τη αρμοδιότητα επιτροπή μα. Ίσως ακολουθήσω κάπως διαφορετική προσέγγιση θα ήθελα σε μια τέτοια ακρόαση όταν μπαίνουμε στις διαπραγματεύσεις του κανονισμού για την επόμενη πολιετή περίοδο να θυμηθούμε ξανά πώς έχουν τα πράγματα. Να φρεσκάρουμε κάπως τις γνώσεις μας. Για την απλούστευση. Προφανώς συμμερίζομαι τα υποθέτα για την απλούστευση διαχειρίσεως των ε, ταμείων πρέπει να εξετάσουμε δύο πτυχές. Πολλές φορές δυσμονούμε μία. Δηλαδή πώς μέσω της διαχείρισης των διεθνωτικών ταμείων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου υπάρχει ε, υπάρχουν μαθήματα του αντλήσουμε όσον αφορά την σωστή διακυβέρνηση. Πρέπει να το δείξουμε, να το υπογραμμίσουμε, να το διαδώσουμε, αλλά ισορροπημένα. μια περιφέρεια που γνωρίζω της Ile de France ακόμα και για την Ile de France η χρήση των ιδιωτικών ταμείων θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο. Θα μπορούσε να βελτιώσει τις πρακτικές διακυβερνήσεως που ακολουθούνται και διαχείρισης των δημοσιονομικών που είναι περίπλοκα. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Καταλαβαίνω βέβαια ότι πολλοί φορείς ζητούν απλούστευση. Και πρέπει να λαμβάνει η χώρα στην αρχή τη διαδικασίας. Όταν παρουσιάζονται τα θέματα και στο, στην περίοδο του ελέγχου. Μεγαλόφωνα σκεπτόμενοι, διερωτώμε, μήπως θα έπρεπε να εμπνευστούμε από αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που έχει τις πιο ριζοσπαστικές και τις περισσότερες αρμοδιότητες και που είναι της μόδα σήμερα σε κάποιες κυβερνήσεις. Δηλαδή στην πολιτική ανταγωνισμού. Διότι εκεί ο καθής γνωρίζει ότι μια από τι σημαντικότερες πτυχέ είναι η διαχείριση των κρατικών ενισχύσεων. Στις κρατικές ενισχύσεις όμως έχουμε τον μηχανισμό de minimis που επιτρέπει αναλογική προσέγγιση στον αφορά του ελέγχου και την κινητοποίηση των ενισχύσεων συναρτήσει των διακυβευμένων ποσών. Δεν λέω ότι πρέπει να τα αντιγράψουμε ακριβώς αυτά, αλλά μπορούμε να τα σκεφτούμε. Και κάτι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε. Είναι η αιρεσιμότητα. Έχει δύο πτυχές. Μακροοικονομική, δεν θα τη συζητήσουμε, είπαμε, αλλά και θεματική ρεσιμότητα και συνάρτηση. Θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξή σας πάνω σε αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν έχει αρκετά χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να φάρμα στις πολιτικές. Δεν θα χρησιμεύσει κάτι τέτοιο. Έχουμε μια κατά μέτωπον επίθεση που να κάνουμε. Με πολλούς ε, φορείς και κυρίως με την Επιτροπή των Περιφερειών, σας το λέω. Υπάρχει μια τάση με είναι, λέμε, λένε, μοιράζουμε τα, δίνουμε τα χρήματα και μετά οι περιφέρειες ασχολούνται πώς γίνεται η επιτόπου κατανομή. Εάν το κάνουμε, ακολουθήσουμε την προσέγγιση, θα πετύχουμε ποτέ στρατηγική. Προσωπικά είναι αυτά που λέω, δεν σμεύω κανέναν. Ούτε εκμεταλλεύουν θέση μας Πρόεδρου. Τα φύγω αυτά, διότι στο Κοινοβούλιο πιστεύω και έναν του Συμβουλίου πρέπει να έχουμε στεναρή θέση. Αλλιώς θα μπούμε σε λογική αποτυχίες και δεν θα πετύχουμε τίποτα. Ακούω και το φίλο μου του Ντελμπάρ τη περιφέρεια που μου λένε ότι η Επιτροπή των Περιφερειών ε, τα γνωρίζει αυτά. Οι περιφέρειες ξέρουν τι ανάγκε του. Ε, λοιπόν, μπορούμε να καταπολεμήσουμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκό την ένδια κλπ. ενοχλούμε. Όταν ξεκινήσαμε τις συζητήσεις, συζήτησα με την κυρία Σουέτερ το θέμα, μία από τις εμπειρογνώμονές μας. Και είπαμε δεν πρέπει να γίνει αυτόνομο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Χρειάζεται ένας κοινό κανονισμός και μετά τα κανονίζουμε μεταξύ μας. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έχουμε μεγάλο κοινό κείμενο που περιέχει τα πάντα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μικρούλι, σημαντικό αλλά μικρούλι. Βλέποντας την περίοδο από την οποία βγαίνουμε τώρα, τι προσπαθείς να κάνουμε. Το 2009 είπαμε ότι χρειάζεται ένα σχέδιο ανάκαμψης. Και τι έχουμε σαν ευρωπαϊκά Γαλλίο γι' αυτό, τα ιδιωτικά ταμεία. Χρειάστηκε να επανεφεύρουμε κάτι που δεν λειτουργήσε σωστά για να πετύχουμε την ευελιξία. Καλό να έχουμε πολιετή συμβάσεις που να υπάρχει νομική ορατότητα κλπ. και να διαρκούν πέντε χρόνια. Αλλά πώς γίνεται η συγκυριακή ε, προσαρμογή. Έχουμε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πουθενά δεν υπάρχει δημιουργία ενός ε, του Ταμείου Συγκυριακής Προσαρμογής. Αν δεν υπάρχει αυτό το εργαλείο, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον ευρωπαϊκό προπλογισμό, πώς θα πετύχουμε τους στόχους εφαρμόζουμε κάποιου κανονισμού που περιμένουμε αποκατάσταση του ευρώ σε 15 χρόνια για να κάνουμε αυτά που θέλουμε και να ρυθμίσουμε αυτό το θέμα. Τέταρτον, τι κάνουμε με τα χρήματα που δεν χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη. Τε, τελευταίο ερώτημα. εταιρική σχέση. Εγώ 100% συμφωνώ μαζί σα. Ποια είναι η δυσκολία. Βλέπω την ισότητα μεταξύ των κρατών μελών. Έτσι τα κράτη-μέλη όπου εκεί που πηγαίνουν τα πράγματα πηγαίνει πάντα καλύτερη η κατάσταση, εκεί που δεν πηγαίνουν τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά, υπάρχουν πολλά προβλήματα και έχουμε δυσκολία να βγούμε από το τέλμα. Η χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε τι θα μπορούσε να συμβάλλει, πώς θα μπορούσε να βελτιώσει τις δομές εταιρική σχέση εκεί όπου αυτές ε, είναι απογοητευτικές. Ενώ όσον αφορά τη σύγχρονη διαχείριση έχουμε δοθεί διακυβέρνηση, έχουμε τη βαθμολόγηση κλπ. Ε, και θέματα να τα εφαρμόσουμε αυτά ή τα χρειαζόμαστε. Θα σας δώσω το λόγο. Ο κύριο Κόνι Ρόιτερ έπρεπε να φύγει. Σίγουρα θα έχουμε και άλλες δυνατότητες να μιλήσουμε μαζί του. Προτείνω να ακολουθήσουμε την αντίστροφη σειρά τη αρχικής σειρά αν συμφωνείτε. ξεκινώντα από την κυρία Jones του APN. UAPN. Σύντομα όμως, ε. Ξέρω ότι είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνετε αυτό, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε ρεαλισμό. Λοιπόν, πέντε λεπτά αν μπορείτε να πάρετε το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Τζόμς. Είναι πάρα πολλά τα σημεία τα οποία ηγέθησαν και είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω σε όλα. Θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της επιστημιστικής βοήθειας, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για το δίκτυό μας. Νομίζω ότι το όλο θέμα είναι λένε πολλοί ότι είναι μη ρεαλιστικό. Πάντα στο παρελθόν είχε χρηματοδοτηθεί από χωριστό κονδύλιο την κοινή αγροτική πολιτική. Το να φέρουμε λοιπόν στο, στα διαδοτικά ταμεία ένα τέτοιο κονδύλιο ότι αυτό θα μειώσει και τα πραγματικά διαθέσιμα χρήματα για τα σχέδια υποστήριξης της κοινωνικής συμπερίληψης και για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πάνε σε θέσεις απασχόλησης ποιότητας. Εάν θέλετε να το κρατήσετε μέσα, τότε πρέπει να αυξήσετε το ποσό της χρηματοδότησης, γιατί το κονδύλιο αυτό ήταν πάντα χρηματοδοτούμενο από άλλους, ε, σε άλλες επικεφαλίδες για την επικέντρωση σε ορισμένους τομείς. Αυτό είναι δύσκολο γιατί από τη μια πλευρά εμείς υποστηρίζουμε τη γενική ευθυγράμμιση με τους στόχους της Ευρώπης 2020, αλλά αυτό θα είναι μόνο αυτό θα είναι πράγματι πολύ περιορισμένο και θα, υποσκάψει τη δυνατότητα ευρύτερη κοινωνική προσέγγιση. Εμεί υποστηρίζουμε μια ευρύτερη προσέγγιση. Πρέπει να κάνουμε σαφέ ποιο είναι ο γενικότερο στόχο, η εξάρτηση τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε μονάχα τα θέματα απασχόληση και κατάρτισης. Αυτά από μόνα τους δεν θα την ένδια. Δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας. Δεν μπορούμε να είναι ρεαλιστικό να φανταζόμαστε ότι όλοι οι απόκληροι θα βρουν μια θέση κάποια στιγμή. Χρειάζεται καλύτερη συμμετοχή σε κοινωνικό επίπεδο και καλύτερη βελτίωση των συνδικών διαβίωσης και υγείας των ατόμων αυτών που είναι αποκλεισμένοι. Για την κοινωνική καινοτομία νομίζω ότι και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και εδώ όμως θα πρέπει να έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι μπορεί να είναι το σύνθημα της ε, στιγμής, αλλά για πολλούς αυτό είναι ο κωδικός για την περικοπή των, ε, ε, υπηρεσιών, για την εξοικονόμηση από τις υπηρεσίες. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι λειτουργεί και να το υποστηρίξουμε και να υποστηρίξουμε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ως την πραγματική βάση για να εξασφαλίσουμε την κοινωνική συμπερίληψη. Αυτό πρέπει να είναι από τα κέρια επιχειρήματά μας για την ε, οικονομική διαχείριση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να ξεπεράσουμε παραγωγικά χάρη το πρόβλημα της καθυστέρησης πληρωμών. Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγικά χάρη προχρηματοδότησης. Να υπάρχει καλύτερη χρήση των συνολικών χορηγήσεων. Όλα αυτά είναι πρακτικά θέματα τα οποία ισχύουν σε πολλές χώρες. Έχουμε καλές πρακτικές. Θα πρέπει αυτές οι πρακτικές να γίνουν στις πρακτικές και να ενσωματωθούν στου κανονισμούς για το θέμα της εταιρική σχέσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δύο πράγματα. Από τη μία πλευρά πρέπει να έχουμε διαβούλευση με τους εταίρους, είτε είναι κοινωνική εταιρεία είτε κοινωνία των πολιτών, για να έχουμε ανάπτυξη ενός κώδικα συμπεριφοράς. Και αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς θα πρέπει να είναι ένα πλήρες έγγραφο, ένα έγγραφο που περιλαμβάνει και παραδείγματα και πραγματικές κατευθυντήριες γραμμές με ε, Παραδείγματος χάρη στην, ε, στους, υπήρχε το εγχειρίδιο που εξέδωσε η Κομισιόν για τις κοινωνικές πτυχές των δημοσίων διαγωνισμών. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει παρακολούθηση, οι κατάλληλοι και σύνδεση με τη στρατηγική 2020 όπου έχουμε την αιτιολογική σκέψη 16 για τις ενσωματωμένες κατερνητές γραμμές. Και πρέπει να βοηθήσει και στην μεταρρύθμιση των εθνικών προγραμμάτων, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα θέμα mainstreaming για να εξασφαλίσουμε την εταιρική σχέση σε όλες τις προοπτικές και πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή πολιτική και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ τα μάλα για το ΣΕΠΕ, ο κύριος Δαβίδ Ανσιό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά σημεία αναφέρθηκαν. Είναι πολύ δύσκολο απαντήσω σε όλα τα μέλη θα χαρώ πολύ να ε, κρατήσω επαφή μαζί σας και να επανέλθω σε ορισμένα σημεία αργότερα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σημαντικό εργαλείο, ένα δύσκολο εργαλείο που είναι η χάραξη των στρατηγικών Νομίζω ότι στα, για τα εργαλεία τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί είναι απαραίτητο να καταλάβουμε, να καταλάβετε γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν και ποιε είναι οι ιδιαιτερότητε κάθε χώρα και έχουμε μια μεγάλη ε, πολυπικιλία στοιχείων που μπορούμε να πάρουμε από του ε, πυρογνώμε. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε μια ανεπαρκή χρησιμοποίηση. Πολλέ φορέ δεν υπάρχουν γνώσει, στα κράτη-μέλη, πολλέ φορέ για το Ταμείο συνοχή, υπάρχουν μονάχα κεντρικοί φορεί οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν το Ταμείο συνοχή αλλά δεν υπάρχει ε, περιφερειακή γνώση. Ενώ σε άλλες χώρες υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει ευρύτερη γνώση και όχι απλώς μια επιχείρηση να λέει «Α, τι ωραίο ψητό θα ζητήσω και εγώ χρηματοδότηση». Υπάρχει επίσης το θέμα της πολυπλοκότητας των ε, αιτήσεων που αποτελεί ένα πρόσκομα. Η ιδέα του de minimis, του συστήματος de minimis, μπορεί να είναι επωφελής. Να απλοποιήσουμε και τα πρότυπα τον χρόνο διεκπαιδεύσης. Η απλοποίηση λοιπόν μπορεί να βοηθήσει όλες τις επιχειρήσεις γιατί δεν έχουν όλοι οι φορείς και οι επιχειρήσεις τις πόρους για να αποκτήσουν την κατάλληλη τεχνογνωσία για να συμμετέχουν στις διαδικασίες που απαιτούνται τώρα. και σχετικά με τα θέματα αυτά τίθεται και το θέμα των εταιρικών σχέσεων, όπως έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, είναι ένα κέριο θέμα. Και επίσης και είναι σημαντική και η χρηματοδότηση για να εξασφαλίσουμε ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα και θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε μια επόφελη συνεργασία μαζί σας και θα σας στείλουμε πραγματιστικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε για το ΕΑΠΕΜ η αρμόδια κυρία. Ευχαριστώ κυρία μου. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα είπατε και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Σας ευχαριστούμε. Έχουν τεθεί συγκεκριμένα ερωτήματα, θα τα απαντήσουμε και εμεί συγκεκριμένα καθώς και θα σας στείλουμε και τις γενικές μας θέσεις. Τρία σύντομα σχόλια για την απλοποίηση θα ήθελα να πω ότι για μας Το θέμα είναι ποια πτυχή της απλοποίησης πρέπει να διαλέξουμε. Κάναμε μια μελέτη για τη συνοχή στις χώρες μέλη και προτείναμε ορισμένα μέτρα απλοποίησης. Ε, παράδειγμα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλη γραφειοκρατία και δεν έχουν το προσωπικό που απαιτείται για να διεκπαιρεώσουν όλα αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό χρειάζεται απλοποίηση. Αν θέλετε να σας πω κι άλλα. Δεύτερον, πολύ ενδιαφέρον, η καινοτόμα λέει οργάνωση της βελτίωσης των πυροσόντων. Το θέμα είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες, στις πραγματικές ανάγκες. Να δούμε τι λείπει για να επιστρέψει κανείς στην αγορά εργασίας, είτε είναι ειδικευμένο είτε είναι ανειδίκευτος ή ανειδίκευτη. Πολύ ενδιαφέρον θέμα πάντως. Τέλος, για τις εταιρικές σχέσεις Πάλι πρέπει να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστούν επιτόπου στην πραγματικότητα. Εμείς... Ε, έχουμε στοιχεία και προσπαθούμε να τα αναλύσουμε. Αυτές οι οργανώσεις που αποτελούν την, τις οποίες αντιπροσωπεύουμε μάλλον θα συνεργαστούν με τα χαράς σε οποιοδήποτε τέτοιο. Στο. Merci beaucoup. Finalement, personne n'avait besoin de 5 minutes, donc c'est parfait. Κανείς δεν χρειάστηκε πέντε λεπτά, τέλεια. Λοιπόν, για την Ευρωπαϊκή ΓΕΣΕ. Εγώ θα χρειαστώ πάνω από 5 λεπτά. Πάνω. Καταρχήν θέσατε τον δάκτυλον επί του τύπου των ύλων, δηλαδή την καλύτερη, και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των δαμείων, αλλά και με καλή διαχείριση, governance. Και ως μέλος μιας οργάνωσης που τη διαχειρίζεται η Τριμερής Επιτροπή του Κοινωνικού Ταμείου. Θα ήθελα να πω ότι μία πρόταση για ένα νέο, μια νέα έτσι τριμερή επιτροπή για καλύτερη διαχείριση governance ή για να συμμετέχουμε και εμείς στις αξιολογήσεις ή monitoring που λέμε αλλά και ex post και ex post έλεγχο. Σωστά τονίσατε ότι το Συμβούλιο πρέπει να αντιμετωπίσει επιγόντως την κρίση και τις επιπτώσεις της που είναι κρίσιμες και δραματικές και αποφάσισε πριν από δύο χρόνια αφού το κοινωνικό ταμείο, να γίνει το κοινωνικό ταμείο ένα από τα εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στην Επιτροπή αυτή διαχείριση του κοινωνικού ταμείου θα έλεγα ότι ακόμη και σε περίπτωση απλοποίησης και ευελιξίας τα ταμεία δεν χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο ούτε καλύτερα. Αντίθετα, υπήρξαν μπλοκαρίσματα. Δεν πρέπει να περιμένουμε λοιπόν την επόμενη προγραμματική περίοδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το μόνο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και η εφαρμογή του κοινωνικού προγράμματος της κοινωνικής πολιτικής που λέγαμε παλαιότερα πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλύτερα. Τώρα, δικαιολογίες που μας δίνουν οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων είναι «Μα είναι πολύπλοκα αυτά πράγματα, είναι συγχρηματοδοτούμενα, έχει γραφειοκρατία». Μα ειναι πολύ αυτα πραγματα ξέρουμε ότι τα διοικητικά είναι πάντοτε γραφειοκρατικά και καθυστερούν. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να βασιζόμαστε σε πολιτικά οράματα και κυρίως σε πολιτική θέληση. Η Ελλάς παραδείγματος χάρη. Δεν χρησιμοποιήθηκε ακόμα για την Ελλάδα το κοινωνικό ταμείο για να βοηθήσει τη χώρα αυτή να βγει από την κόλαση στην οποία βρίσκεται. Πορτογαλία, Ισπανία, άλλοι κτλ. Τα ίδια. Και εδώ έτσι απαντάω εν μέρη τουλάχιστον στο ερώτημά σας τι να κάνουμε. Εμείς ήδη είπαμε και το δέχτηκαν αυτό και μερικοί ευρωβουλευτές να χρησιμοποιηθεί περισσότερο το κοινωνικό ταμείο. Όταν λύγει μια προγραμματική περίοδος εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και μπορούμε εκεί να προσθέσουμε μια ποσόστοση, ένα ποσοστό για να βοηθηθούν οι χώρες αυτές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες να βγουν από την κρίση. Και σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει ακόμα και στα γαλλικά μια task force έχουμε για την Ελλάδα. Έτσι κάνουμε εμείς οι συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες. Άρα με συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων και των συνδικάτων. Επομένως τελικά σκεφτείτε το κυρία Πρόεδρε. Καλύτερη χρησιμοποίηση ενός ταμείου συγκυριακής προσαρμογής αφού υπάρχει ταμείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση γιατί όχι και αυτό. Άλλο ερώτημα. Για μας η θεματική οργάνωση και συγκέντρωση είναι κάτι που μπορούμε να το δεχτούμε αλλά ακόμη καλύτερα αν συμμετέχουμε περισσότερο στον καθορισμό του κοινού στρατηγικού πλαισιού που θα οριστεί και ενωσιακά και εθνικά και περιφερειακά και τοπικά. Αλλά με συνέπεια και συνοχή. Μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε προτεραιότητες και θεματικές ομάδες και για τους πόρους. Αλλά για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που ευτυχώς επέζησε γιατί είχε συζητηθεί και στην περίληψή του σε άλλα και άρα κατάργησή του πρέπει να συγκεντρωθεί όχι να προσθεθούν άλλα ταμεία όπως βοηθεία στους πιο στους πτωχοτέρους Αυξήθηκαν μεν τα κονδύλια του, αλλά, αλλά άμα αφαιρέσουμε τις προσθήκες, πού καταλήγουμε, πουθενά. διατηρούμε τα υπάρχοντα εργαλεία όπως το πρόγραμμα βοήθειας για τους υποδεέστερους είναι σε πλήρη αντίφαση με την απόφαση να καταργηθεί ενώ αυξάνεται η ανέχεια. Παρακαλώ μπορείτε να τελειώνετε λέει πρώτα. Ναι, ναι, τελειώνω ήδη. Λοιπόν, το άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι η σημασία των παρατηρητηρίων. Λέτε πρέπει να υπάρξουν προβλέψεις, προοπτικές. Έτσι λέτε. Άρα για να γίνουν οι προβλέψεις χρειάζονται και επιχειρήσεις που να τις κάνουν. Υπάρχουν ήδη παρατηρητήρια για την απασχόληση περιφερειακά, τοπικά και πρέπει και αυτά να συνδυαστούν μεταξύ τους. Η κυρία η σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα όλες τις παρεμβάσεις και τις ερωτήσεις που ετέθησαν, τις απαντήσεις των εταίρων μας με τους οποίους συνεργαζόμαστε τακτικά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία που θεωρώ ουσιοδέστατα. Πρώτον, συμφωνούμε, θεωρώ, επί της αναγκαίας συγκεντρώσεως επί των στόχων. Πολιτική ευρωπαϊκή της απασχόλησης πρέπει να επικεντρώνεται επί της εντάξεως της επαγγελματικής, πρώτα απ' όλα, Νομίζω ότι αυτό είναι θεμελιώδη σημασία. Πολλοί από εσά το αναφέρατε. Το είπαν οι εταίροι μας που μίλησαν το πρωί και οι βουλευτέ. όπως ο Τόμας Μαν. Η συγκέντρωση για μας πρέπει να είναι υποχρέωση και ε, ένας πύχη Αυτό προσπαθούμε. Στους στόχους ανέφερε κάποιος η κυρία Τζόνς. απειλούνται και απειλείται και το 20% για την πολιτική της αλληλεγγύης και καταπολέμηση της ένδυας. Συζητείται στο Συμβούλιο αυτό και θα πρέπει να κινητοποιηθούμε όσον αφορά αυτό το θέμα. Δεύτερον, αποτελεσματικότητα, αυτή που επιδιώκουμε όλοι. Αρκετοί το ανέφεραν το θέμα. Θέλω να στραφώ προς εταίρους μας, για να πω κάτι. Ε, στόχος μας είναι ένα κοινό δύσκολο. Χρειάζονται συγκεκριμένες μέθοδοι εργασίας. Κατά περίπτωση μέθοδοι. Το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε ε, χρειάζεται να γίνεται προσμέτρηση να εντοπίσουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν και κάποιες ομάδες που ξεφεύγουν από την γενική πολιτική. Γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία με του εταίρους. Είναι πάρα πολύ σημαντική συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, με συνδικάτα, οργανώσεις, ε, μη κυβερνητικές κλπ. Δεν μιλάμε για τη μάζα, έχουμε μπει στη λεπτομέρεια. Και αν θέλουμε αποτελεσματικότητα, χρειάζονται συγκεκριμένες λύσεις ειδικέ για τις διάφορες ομάδες που θέλουμε να καλύψουμε. Τρίτον, πρόβλεψη. Το είπανε τα συνδικάτα και οι ενώσεις. Και οι βουλευτέ. Και δεν είναι κάτι εύκολο αυτό. Υπάρχουν φορείς διάφοροι για αυτό το θέμα. Με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ αυτό κουβεντιάζαμε για την επαγγελματική κατάθεση πώς μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, ούτως ώστε να γίνεται σωστή ένταξη επαγγελματική εκείνων που, είναι στο, που είναι στο περιθώριο σήμερα. Χρειάζεται πολλή δουλειά να κάνουμε για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Πρέπει να πω ότι σήμερα δεν είναι εύκολη η κινητοποίηση του κόσμου του επιχειρηματικού και του διοικητικού προβλέποντας τι θα γίνει στο μέλλον. Χρειαζόμαστε ευελιξία, αλλά έχουμε και στόχο μέχρι το 2020 όλοι απέναντί μας κινούνται βραχυπρόθεσμα. Άρα πρέπει να αλλάξει αυτό και να προχωρήσουν πιο πέρα οι προθεσμίες. Τέταρτον, για το πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας προς τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και την ένταξη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Άκουσα αυτά που είπατε. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι στο κανονισμό πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αντικατοπτρίζεται ως ποσοστό τον Ταμείο Συνοχής. 40% το Ταμείο Συνοχής προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας Δυσδύει στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το λέτε, εντάσσεται εκεί. Αλλά είναι δύσκολο έτσι που υπάρχει γενική προσέγγιση να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Χρήση των πόρων. Είδα τι γίνεται σε πολλές χώρες και σε πολλές περιοχές όσον αφορά τη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αρχές 2012 είμαστε. Το πρόγραμμα αυτό λύγει το 2013, τα προγράμματα. Έχουν καταβληθεί το 30% των πόρων. Έχουμε 30% που έχουν δεσμευτεί για προγράμματα που θα ολοκληρωθούν το 2013. Μας μένει το 1 τρίτο περίπου των πόρων που θα έπρεπε κανονικά να υποστηρίξει προγράμματα που θα ξεκινήσουν τώρα για να λήξει το 2013. Υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν όσον αφορά την επεξεργασία των προγραμμάτων και πρέπει να κάνουμε πολλές προσπάθειες. Όλοι μαζί τους ώστε αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιηθούν να υπάρξει εταιρική σχέση σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται αυτή η εταιρική σχέση. Και τέλος κυρία Πρόεδρε, 300% συμφωνώ με την ανάλυση σας όσον αφορά την συνοχή που χρειάζεται να υπάρχει μεταξύ ευρωπαϊκών πολιτικών και της τοπικής εφαρμογής αυτών. Ξέρω πόσο οι περιφέρειες είναι λέμαργες. Ναι, Θέλουν να έχουν στα χέρια τους ευρωπαϊκά χρήματα για να εφαρμόζουν τοπική πολιτική. Αν θέλουμε να κερδίσουμε τη μάχη της απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μας χρειαστεί στεναρή στάση. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Τέλειωσε αυτό το τμήμα. Τις επόμενες ημέρες θα καταθέσετε φαντάζομαι το έγγραφό σας και τα λοιπά. Τώρα το 26. Ευχαριστώ τους δύο υποψηφίους για τη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕΕ. Με μεγάλη χαρά βλέπω τον προκάτοχό μου. Όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορίζει τρία μέλη του στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Και προηγουμένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ορίσει κατά την πρώτη περίοδο τρία μέλη, την κυρία Σαραπάρκη, τον κύριο Σανφρασουά Μεζιέρ και τον κύριο Χριστόπουλο. Χρειάζεται τώρα να ακούσουμε τους δύο υποψηφίους που είναι εδώ και προτείνω πρώτα να ακούσουμε τον απερχόμενο Ζαν Φρανσουά Μεζιέρ που μας είπε ότι είναι διαθέσιμος να ξαναπάρει την ίδια θέση και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Ιαν Άντερσεν. Κύριε Ιωάννη Φραγκίσκο Μεζιέρ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ να μας πείτε και γιατί θέλετε να ανανεώσετε τη θέση σας και ποιο είναι το όραμά σας αφού έχετε εμπειρία εκεί. Ευχαριστώ Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Εγώ θέλω να θέσω και πάλι υποψηφιότητα για τρεις λόγους, πολύ απλά. Πρώτα απ' όλα, όπως αναφέρατε, ο κανονισμός ο οποίος διέπει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την ε, κατάρτιση έχει τροποποιηθεί το Δεκέμβριο του 2008. Μετά από τρία χρόνια μπορούμε να κατανοήσουμε ότι δίδει πολύ σημαντικές και εύστοχες αποστολές στον φορέα αυτό. Καταρχήν από μια γενική έποψη για την παροχή πληροφοριών σε σχέση με την ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Και αυτό είναι ένα σημαντικό διακυβευόμενο σε χώρες που είναι σε ταξιακή φάση και στις χώρες της γειτονίας Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν και ιδίω για τις χώρες ε, της γειτονίας μας στην νότια όχθη της Ευρώπης, του Μαγκρέ που είναι δημοκρατικής παράδοσης. Εκεί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων που είναι σημαντικό στόχος του Ιδρύματός μας. Δεύτερον, εδώ και τρία χρόνια έχει κινητοποιηθεί ιδιαίτερα το ο φορέας κατάρτισης για να αντιμετωπίσει τα διακυβευόμενα αυτά που αναφέρατε. Πιστεύω ότι έχει πράγματι μια πραγματική εμπειρογνωμοσύνη και την οποία την αναγνωρίζουν και οι χρηματοδότες και οι χορηγοί. Χωρίς λοιπόν να χρηματοδοτεί έχει την εμπειρογνωμοσύνη το Ίδρυμα αυτό και την χάνει αυτή η λειτουργία του αναγνώρισης και άμεσης πρόσβασης στους υψηλούς πολιτικούς κύκλους. Αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμο επίσης το Ταμείο, το Ίδρυμα αυτό γνωρίζει και τη σχέση μεταξύ των εσωτερικών διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδικασία της Κοπενχάγης και τις ε, ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στις χώρες γειτονίας και έχει εργαστεί ιδιαίτερα στα ουσιαστικά στοιχεία αυτής της συνεργασίας. Κατά κάποιον λόγον λοιπόν, κατά κάποιον τρόπο, εδώ και τρία χρόνια, έχει αναπτύξει νέες εταιρικέ σχέσεις το Ίδρυμα αυτό, <clears throat> έχει ανανεώσει τις ενεργειές του και νομίζω ότι είναι ανεγνωρισμένη η εμπειρογνωμοσύνη του. Τρίτο στοιχείο, μαζί με τους συναδέλφους μου, την Σαραπαρκίν, η οποία θέλει να συνεχίσει το έργο αυτό, προσπαθήσαμε να βρούμε τη σωστή η ισορροπία με το να τακτικές ε, εκθέσεις στην Επιτροπή σας, να συναντούμε τους κοινοβουλευτικούς που θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Όλα αυτά είναι σημαντική επένδυση και θέλω λοιπόν να τονίσω τη σημασία αυτής της επένδυσης προσωπικά. Εγώ είμαι ειδικό στους ανθρώπινους πόρους και στην κατάρτιση. Υπήρξα επικεφαλής της ε, των υπηρεσιών κατάρτισης μιας γαλλικής περιφέρειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει και σας βέβαια. Αυτό είναι χωριστό θέμα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα θέματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί είχα εκλεγεί πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική κατάρτιση, ένα από τα σημαντικότερα δίκτυα στον τομέα αυτό, που έχει σε στόχο την παγκόσμια αναγνώριση για την γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη του. Αυτά λοιπόν κυρία Πρόεδρε, για όλους αυτούς τους παρατεθέντες λόγους θέλω να ανανεώσω τη θητεία μου, ώστε να υπηρετήσω το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε να ακούσουμε τους άλλους υποψηφίους και μετά να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, αν θέλουν τα μέλη να θέσουν ερωτήσεις. Αγαπητέ συνάδελφοι, είναι χαρά να σας δίνω το λόγο και να έχω τη δυνατότητα να σας χαιρετήσω σε αυτή την αίθουσα. Μου είπατε ότι είστε διαθέσιμος να απαντήσετε σε ερωτήσεις των συντονιστών, να είσαστε υποψήφιος. Γιατί θέλετε να είστε υποψήφιος. Πώς βλέπετε αυτό το καθήκον σας έχοντας, ε, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχετε στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ που ε, Χαίρομαι που επέστρεψα και βλέπω τους παλιούς μου συναδέλφους. Τόσα χρόνια πέρασαμε μαζί. 14,5 χρόνια ήμουν εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν επέστρεψα έκτοτε εδώ και τρία χρόνια έφυγα. Το Μάιο Θάρο, του 2009. Και μετά ήμουν στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο, μήνα Ιούλιο τότε. Και ήταν η τελευταία μου φορά τότε που ήμουν στο Κοινοβούλιο. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που επιστρέφω. Πρώτα απ' όλα να πω κάποια πράγματα για την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο είναι ένα σημαντικό θεσμικό όργανο, αλλά για μένα ήταν και ένα πανεπιστήμιο. Μαθαίνεις πολλά κατά τη διάρκεια της θητείας σου εδώ. Σωρεύεις γνώση σαν πανεπιστήμιο είναι. Το λέω σε πολλούς στη Σουηδία. Τους μιλάω για τη δουλειά που γίνεται στο κοινοβούλιο. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειε για το Ίδρυμα. Το ξέρω, αλλά κάποια γενικά σχόλια να πω και γιατί θέλω να είμαι υποψήφιος. Τα γενικά μου σχόλια αφορούν τις προκλήσεις. Ποιες είναι οι προκλήσεις για την Ευρώπη. Το κουβεντιάσατε σήμερα. Α, δεν αναφέρομαι συχνά σε προβλήματα. Μιλώ για προκλήσεις. Καλύτερα έτσι. Βλέπεις μπροστά σου προπτικές. μπορεί να τα λύσεις. Τα προβλήματα είναι πιο δύσκολα. Η οικονομία, η ανάπτυξη, η ανεργία, αυτά είναι οι προκλήσεις. Ποσοστά απασχολησιμότητας και τα κοινωνικά θέματα, ε, και πώς σηματοδοτούνται τα συστήματα πρόνοιας. Σε κάποιες χώρες οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες. Αλλά υπάρχουν για κάθε χώρα. Όταν έφυγα από το κοινοβούλιο, παρέμεινα δραστήριος. Στο βιογραφικό μου λησμόνησα ότι δούλεψα σαν δάσκαλος από 16 χρόνια, από το 72 μέχρι το 88. Ακούγοντας την κουβέντα για το κοινωνικό ταμείο ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σουηδικού Κοινωνικού ε, Ταμείου. Δεν υπάρχει πλέον Διοικητικό Συμβούλιο. Τότε όμως ήμουνα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μία από τις βασικές προκλήσεις είναι η παιδεία. Έτσι νομίζω. Ε, ε, είμαι στο Χέλσιμπορ, στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι υπεύθυνο για την παιδεία. Βλέποντα τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Και εκεί υπάρχει ανεργία. Και εμείς έχουμε ανεργία. Και να, ανισότητες. βλέποντα τους ανέργους σήμερα. Βλέπουμε ότι είναι οι νέοι. Αλλά όχι όλοι. Είναι οι νέοι εκείνοι που δεν έχουν ε, κατάλληλη παιδεία. Αυτοί που έφυγαν νωρί από το σχολείο τους λείπει παιδεία. Δεν βλέπει συχνά ανεργούς νέους με εκπαίδευση. Καμιά φορά το αν έχουν πάρει λάθος πτυχίο, αλλά όχι τόσο συχνά. Αν δούμε το έτσι 45, 50, 55 και σε μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και με λάθος ε, εκπαίδευση. Τι πρέπει να κάνουμε. Επανειλημμένα το συζητήσαμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα εκπαιδευτικό για όλους, για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ποτέ δεν είναι αργά. Οι νέοι πρέπει να έχουν δεύτερη, τρίτη ευκαιρία, τέταρτη ευκαιρία για να πετύχουν σωστή παιδεία. And for, Για τους ηλικιωμένους Παιδεία. Εκπαίδευση. Ακόμα και εγώ. Είμαι 64 τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Αυτές είναι οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ίδρυμα Κατάρτισης αφορά τις γειτονικές χώρες, τις χώρες εταίρους. Κάποιες θα γίνουν μελλοντικά μέλη της Ενώσεως. Άλλες χώρες είναι εταίροι. Και ερχόμαστε συχνά σε επαφή μαζί τους. Είναι σημαντικό και για μας. Πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά συστήματα, να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι σε αυτά και να αναπτυχθούν εκπαιδευτικά συστήματα σωστά με αυτή τη συμμετοχή στις άλλες χώρες. Μιλώντας για τη Βόρεια Αφρική. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το σύστημα πρόνοιας και η παιδεία. Ε, το πρόβλημα είναι και η δημοκρατία. Αν θέλουμε να αναπτυχθούν αυτές οι χώρες, να είναι καλή εταίροι για μας, επιτυχής εταίροι, αυτό θα κάνει καλό και σε εμά. Αν το θέλουμε αυτό λοιπόν, πρέπει και αυτοί να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά συστήματα και συστήματα για διαβίου εκμάθηση. Και να μπορεί ο νέος να βρίσκει δουλειά και ούτω καθεξής. Έτσι θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, θα υπάρχει ε, ε, σωστή ε, απασχόληση, παγίωση της δημοκρατίας, εποφελές για όλους. Και για εκείνους και για μας. Χάρη κατά μάλα όταν μου ετέθη το ερώτημα. Τα μάλα σα λέω. Όχι μόνο να υπάρχει σχέση με να έχω επαφή με την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο που την αγαπώ τόσο μετά από 14,5 χρόνια. Όχι μόνο γι' αυτό, δεν χάρηκα μόνο γι' αυτό. Αλλά χάρηκα που ετέθησα όλε τις διαστάσεις, η ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά και άλλη διάσταση τη περιοχή μου. Που δεν είναι στην Νότια Σουηδία, αλλά είναι κοντά και στη Δανία με την Κοπενχάγη, 50 χιλιόμετρα από την Κοπεχάγη είμαστε. Μια γειτονιά είμαστε, ίδια αγορά εργασία. Και προσβλέπω την συμμετοχή μου στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης και προσβλέπω και σε μελλοντικέ επαφές μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Στρέφομαι προς τους συναδέλφους αν θέλει κάποιος να θέσει ερωτήματα στους υποψηφίους. Κύριε Θέρκας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι πραγματικά ένα ερώτημα. Απλώς θα ήθελα εξ ονόματος των σοσιαλιστών συναδέλφων θα ήθελα να εκφράσω την αυροφροσύνη μας προς τους υποψηφίους και στο τρίτο υποψήφιο που το γνωρίζουμε μονάχα από την έγγραφη υποβολή του. Θέλω να σας ε, διαβεβαιώσω ότι θα έχετε τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής αυτής. Ο κύριος Μεζέρ ξέρει ότι εξετάσαμε το βιογραφικό του στην συνεδρίαση των συντονιστών και βλέπουμε τώρα ότι πράγματι τον αδικεί το βιογραφικό του και ελπίζω λοιπόν ότι θα είναι μια ε, επιτυχής ε, θητεία, αλλά κυρίως θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής μας αυτόν τον κύριο Άντερσεν. Νομίζω ότι έχω εργαστεί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί του και τώρα βλέπω ότι εξακολουθεί να μένει νέος και σφρίγιλος και πάντα δεσμευμένος με την Ευρώπη. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τους νέους και έχει βελτιώσει και την ακαδημαϊκή του ε, παιδεία, αλλά έχει παραμείνει δεσμευμένος και προσιλωμένος στην πράξη να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Είναι μια πολύ καλή υποψηφιότητα και η εμπειρογνωμοσύνη του μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας. Αγαπητέ Γιάν, θα δουλέψουμε πολύ καλά μαζί. Καλώς ήρθες στο ίδιο στο σπίτι. Και θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να σας πω ότι αν υπάρχουν μόνο τρεις υποψήφοι για τρεις θέσεις, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που είχαμε αποφασίσει χθες να μπορούμε ίσως διαβοής να εγκρίνουμε και τους τρεις υποψηφίους εάν συμφωνείτε. Σας ευχαριστώ οι συντονιστές του, ο συντονιστής του ΕΡΚ έθεσε το θέμα αυτό ήδη στη μέση διάταξη αλλά δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο. Όταν έρθει κατάλληλη στιγμή θα αντιμετωπίσουμε αυτό το σημείο η κυρία Λαμπέρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τις παρουσιάσεις που μόλις ακούσαμε. Έχω μερικά ερωτήματα. Οι ορισμοί από το Κοινοβούλιο τι άλλαξαν στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι μία από τις από τους οργανισμούς, από τα ιδρύματα που ασχολούνται με την απασχόληση και γι' αυτό θέλω να μας πείτε και εσείς τι θεωρείτε ότι προσθέτουν οι υποψήφοι για τη διαχείριση του Ιδρύματος ή γενικότερα για το πρόγραμμά του. Κανείς άλλος. Εγώ στο πνεύμα της ερωτήσεως της κυρίας Λαμπέρ θα σας ρωτήσω και τους δύο. Το εξής, το ένα φορά, ερώτημα αφορά την εμπειρία και το άλλο τις προβλέψεις του υποψηφίου. Λοιπόν, αν στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχουν μέλη που ορίστηκαν από το Κοινοβούλιο, με εγγύηση βέβαια της ανεξαρτησίας τους γιατί διάβασα το καταστατικό και τη διαδικασία παρόλα αυτά κάτι μου έχει μείνει στο λαιμό για τα κοινωνικά αν θέλουμε να κερδίσουμε τον αγώνα των ιδεών, μαζί ενώπιον των ηθινόντων στην οικονομική κατάσταση πρέπει και εμείς να έχουμε την ίδια γνώση, την ίδια ικανότητα να αντιπαραβάλουμε τα δεδομένα και να βασιστούμε σε επιστήμη. Όταν από τη μια μεριά εργάζονται οι εμπειρογνώμες και από την άλλη οι πολιτικοί δεν γίνεται τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι οι πολιτικοί θα μας φέρουν τους εμπειρογνώμονες. Αλλά και το αντίθετο είναι δύσκολο. Εγώ έχω γνωρίσει εμπειρογνώμονες που θεωρούν ότι δεν θα δεχτούμε διαταγές από πολιτικούς. Μάλιστα. Πώς όμως θα βεβαιωθούμε ότι τα προγράμματα συμφωνούν χωρίς πολιτική προειδέαση συμφωνούν με τα αποφάσεις στέντα. Στο Τωρίνο αν δεν απατώμε, α όχι στο Δουβλίνο. Στο Δουβλίνο είχα ζητήσει κάποια βοήθεια για τον απολογισμό, κοινωνικό απολογισμό των μέτρων λιτότητας και μου είπανε α όχι. Όχι αυτά είναι της Κομισιόν. Θεωρείτε λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουμε το καταστατικό του Ιδρύματος ώστε να μπορεί να υπάρξει ένας καλύτερος διάλογος. Ή μήπως να ζητήσουμε μελέτη, για να μπορούμε να ζητήσουμε μια μελέτη και τα λοιπά, αν και αυτό δεν είναι μεγάλα, ε, απλώς ερωτώ. Και δεύτερο ερώτημα. Στο πρόγραμμα του Ιδρύματος Κάνετε βέβαια τις μελέτες σας με τη δέουσα επιστημονική ελευθερία, αλλά πώς μπορούμε και εμείς να υποφεληθούμε. Αυτά βέβαια ξεπερνάνε κάπως το πλαίσιο μιας ακρόασης υποψηφίων, αλλά για μας είναι σημαντικό θέμα. Και το είχα πει και σε άλλους διευθυντάς ιδρυμάτων. Θέλετε την ίδια σειρά ή ανάποδα. Την ίδια, την ίδια. κυρία Πρόεδρε. Για το να τροποποιήσουμε το καταστατικό του Ιδρύματος, εγώ δεν το πιστεύω ότι αυτό είναι θετικό. Υπήρξε ένα κείμενο συμβιβαστικό. Αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί και πάλι μια συμβιβαστική λύση αυτού του είδους και όσο έχει το καταστατικό μας επιτρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα. Η επίσκεψη που κάνετε και με άλλους κοινοβουλευτικούς στο Ιδρυμά μας δείχνει ότι όλα τα μέλη του Ιδρύματος είναι έτοιμοι πάντα να ακούσουν τις ερωτήσεις των βουλευτών, επίσημες ή ανεπίσημες, και να δώσουν απάντηση σε ό,τι αφορά την γνωμοσύνη που μπορούμε να προσφέρουμε σε εσά άμεσα. Νομίζω ότι πράγματι το είχα τονίσει ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση υβριδικού χαρακτήρα. Δεν έχουμε σαφή εντολή, είμαστε ανεξάρτητοι, αλλά συγχρόνως με τους συναδέρφους μου προσπαθήσαμε να βρούμε μια ισορροπία και αυτό μπορεί να βελτιωθεί βέβαια τη σωστή ισορροπία γιατί μέσα στο Ίδρυμα πρέπει να έχουμε και ευήκον ους για τις ε, ε αιτήσει του Κοινοβουλίου να παρακολουθούμε τις εργασίες σας και τις προτεραιότητές σας και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι προτεραιότητε του Κοινωνικού Ταμείου για τα θέματα αυτά και επίση με τρόπο συμμετρικό <clears throat> κάνουμε και εμείς εκθέσεις ίσως ε, κάπως ε, πρόχειρου επίπεδου σε σχέση με αυτά που γίνονται με το Ίδρυμα, με τις εκθέσεις που εξετάζονται εκεί κτλ. Είναι σημαντικό λοιπόν στην διεύθυνση του Ιδρύματος να υπογραμμίσω ότι η Κομισιόν ε, σημαντικό ρόλο γιατί αυτή είναι ο εντολέας αλλά εμείς σίγουρα μπορούμε να επηρεάσουμε σημαντικά τις προτεραιότητες της Κομισιόν και εγώ προσωπικά συμμετέσχα σε ομάδες εργασίας η οποία εξεπώνησε το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο εργασίας του Ιδρύματός μας. Επομένως μπορούμε να τονίσουμε ότι υπάρχουν εμπειρογνώμονες στα οικονομικά και στα νομικά, αλλά και εμπειρογνώμονες για τους ανθρώπινους πόρους που γνωρίζουν τη λειτουργία της αγοράς, της εργασίας, της πολιτικές ε, εκπαίδευση και κατάρτισης σε εγκάσιο επίπεδο και που οδηγεί πολλά, σε πολλά διακυβέρματα για τις ε, χώρες που βρισκόνται κοντά στην Ευρώπη, μετακίνηση επιχειρήσεων, μετακίνηση με μεταναστευτικά ρεύματα κτλ. Επομένως, το να μπορεί κανείς να συμμετέχει άμεσα στο έργο του Ιδρύματος αυτού και το να μπορεί να λειτουργεί εκεί. Εγώ προσωπικά είχα λειτουργήσει με την, είχα έρθει σε επαφή με την Ισιακή κυβέρνηση για λογαριασμό του ιδρύματο και μπορούμε με τον τρόπο αυτό να αντλήσουμε πληροφορίε, οι οποίε είναι πάρα πολύ μα. Επομένω δεν πρέπει να τροποποιήσουμε το καταστατικό αλλά να βρούμε τρόπους για να το χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Άντερσεν. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Οι ερωτήσεις της Ζιν Λάμπερτ και της Προέδρου είναι αλληλένδετα. Αν το Ευρωπαϊκό αν κερδίζει κάτι του εμπειρογνώμονε, κάποιοι εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, θα έπρεπε. Κατά κάποιο τρόπο κερδίζει. Αν διορίζεται εμπειρογνώμονε, αν κερδίζεται από το διορισμό ε, εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να διατηρούμε μια σχέση μεταξύ μα. Μπορούμε να συζητούμε μπορώ να παρακολουθώ πώς διεξάγονται οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τις συνδυάσω με τη θέση μου στο Διοικητικό Συμβούλιο και αντιστρόφως. Αυτά που συμβαίνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και οι συζητήσεις εκεί μπορούν να σας διαβιβαστούν και να αντιδράστε εσείς. Κάνουμε τα σωστά πράγματα. Πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν έχουμε δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά μπορούμε πιστεύω να συμβάλλουμε. Αν ενδιαφέρεται κάποιος που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν μπει στο πνεύμα των εργασιών, μπορεί να δραστηριοποιηθεί, να είναι πολύ δραστήριος. Δεν γνωρίζω πολλά για το πρόγραμμα εργασίας, το υφιστάμενο και τι συνέβη. Θα έρθω στα γρήγορα σε επαφή με το ETF και μπορώ σε λίγες μέρες να δω τι κάνουν εκεί στο Ίδρυμα. Να μάθω. Δεν πάρει να λειτουργήσει κανείς σε διοικητικό συμβούλιο αν είναι άσχετος, άμα δεν ξέρει τι τρέχει, πώς είναι το πρόγραμμα. Και όταν τα μάθω αυτά και όταν συνηθίσω τη δουλειά στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα ήθελα πολύ να επανέλθω εδώ και να κουβεντιάσουμε. Τα, τα πάμε καλά, κάνουμε τα σωστά πράγματα. Το Κοινοβούλιο τι θέλει να κάνουμε. Είναι πιο σημαντικά κάποια προγράμματα από άλλα, να ξεκινήσουμε καινούργια μπορούμε να το θέσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να πούμε, κοιτάξτε, αυτό είναι σημαντικό. Α, τέτοιου είδου συζητήσει μπορεί να γίνουν. Εάν διορίσετε εμπειρογνώμους όπως αποκαλούνται, θα έχετε κάποιο όφελος. Πρέπει να υπάρχει επαφή, διασύνδεση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων σας και της Επιτροπής σας. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η σχέση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτήν τη διαθεσιμότητά σας, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των αποφάσεων που πρέπει να πάρουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα να πάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Οι δύο συντονιστές του ΕΛΚ και του S&D μου πρότειναν, προτείνω και εγώ, τα μέλη που διορίσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο να, τα, να ανανεώσουμε την, έτσι απλά την ε, θητεία τους. Έχουμε ένα νέο μέλος και δύο που θέλουν να ανανεώσουν τη θητεία τους. Και τους έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι θα είναι ενεργά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να κάνουν αυτό, τουλάχιστον αυτό που θέλουμε και τους εύχομαι καλή δουλειά εν ονόμετι των μελών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων γνωρίζετε. Μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας θα μεταβεί εις Τωρίνον φέτος στο Τωρίνο και θα έχετε δυνατότητα να το συναντήσετε. Ακόμα και αν δεν είναι μια αντιπροσωπεία της οποίας προεδρεύω. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω. Nous en avons terminé avec ce point. Τελειώσαμε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Ραντεβού στην επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή 13 Φεβρουαρίου στι 7 το απόγευμα στο Στρασβούργο. Γεια σας.